Ε, Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Με συγχωρείτε πολύ που καθυστερήσαμε τόσο πολύ να ξεκινήσουμε, αλλά υπήρχε μια άλλη συνάντηση πριν ταυτόχρονα. Θα αρχίσουμε αμέσως λοιπόν, με συγχωρείτε. Ως προς την ημερήσια διάταξη. Έχουμε διήμερη συνεδρία της Επιτροπής Ήτρε σε τέσσερα τμήματα. Ξεκινάμε λοιπόν. Πρώτο σημείο, έγκριση της ημερήσιας διάταξης υπάρχει στους φακέλους σας. θα το σας ε, έχετε παρατηρήσεις, όχι. Έτσι κι ε, μπορούμε να προσθέσουμε ό,τι θέλετε στα διάφορα. Σημείο 2. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Να θυμίσω σε όλους τους συναδελφούς ότι είστε προσκεκλημένοι στο χριστουγεννιάτικο ποτό μετά τη συνεδρίαση περίπου στις 6.30 μπροστά στην αίθουσα συνεδρίασης. Σήμερα, σήμερα το απόγευμα. Όχι αύριο, γιατί και αύριο το απόγευμα έχουμε συνεδρίαση. Θα ήθελα το χριστιανιάτικο αυτό ποτό να το πιούμε απόψε. Θα είναι και κάποιοι επίτροποι μαζί μας και πρώην επίτροποι επίσης επίτροποι οι οποίοι έχουν συνεργαστεί στενά με την επιτροπή μας. Είναι παλιοί μας φίλοι. Να πω για το σημείο 12 και να σας ενημερώσω ότι αύριο 4 Δεκεμβρίου το απόγευμα τα σημεία 12 και 13 αλλάζουν θέση και το σημείο 12, σχεδιασμό για το Διεθνή Χάρτη Ενέργεια 2015, παρουσίασε από τον Γενικό Γραμματέα του Χάρτη Ενέργεια, δόκτωρα Ούρμπαν Ρουζνάκ. Παίρνει τη θέση του σημείο 13. Έκθεση ιδέε πρωτοβουλία ευκαιρίε πράσινη ανάπτυξη για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αυτά για το αυρενό απόγευμα. Σημείο 3. Έγκριση πρακτικών. 1η και 2 Σεπτεμβρίου, 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 5 και 6 Νοεμβρίου. Όλα τα πρακτικά. Υπάρχουν στην αίθουσα. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μέχρι το τέλος της πρωινής συνεδρίασης. Θεωρούμε ότι είναι εγκεκριμένα τα πρακτικά. Μέχρι τις 12.30 έχετε χρόνο για τις αντιρρήσεις σας ή τις παρατηρήσεις. Σημείο 4. Δημόσια ακρόαση. Υποστήριξη καινοτόμων νεοειδριόμενων ή νεοσύστατων εταιριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μας ενδιαφέρει το τι γίνεται με τις νεοσύστατες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θέμα που το ακούμε εδώ και καιρό και τώρα επιτέλους αρχίζουμε να το μελετάμε και να το επεξεργαζόμαστε με περισσότερη σοβαρότητα. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τους ομιλητές και να τους ευχαριστήσω εξ ονόματος της Επιτροπής Ήτρε που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας. νομίζω θα είναι μια καλή αρχή. Για τη δουλειά μα σε σχέση με τι νοσίστατε επιχειρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε το ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσει αυτέ και οι εταιρείε αυτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίε συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. έχουν ένα ρόλο να διδραματίσουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει στο να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεφύγει από την κρίση. Δικό μα ρόλο λοιπόν είναι μέσα τη έγκριση του κόσμου, του Horizon 2020. Και επιμένοντας να παρακολουθούμε όλες τις δραστηριότητες που ε, έχει αναλάβει η Επιτροπή μας, βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει μια έντονη έμφαση στο ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως το Small Business Act στο Horizon 2020. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα για τις μικρόμεσες επιχειρήσεις για να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια και τις πιστώσεις και να ξεκινήσουν να ε, λειτουργούν από την ε, σκοπιά αυτή είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα COSME. Η πράσινη ανάπτυξη και ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η... ο τίτλος της δικής μας έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας. Η συγητής είναι ο κύριος Ντεμπάκερ. Πολύ σημαντική έκθεση. Και ε, στο τέλος ε, πια της δικής μου εισήγησης, σε ό,τι αφορά την διοργάνωση της ακρόασης, να σας ενημερώσω συνάδελφοι και τους ομιλητές μας ότι προβλέπονται 3,5 ώρες. Δυστυχώς τώρα πια είναι 3 ώρες και 15 λεπτά. Αυτό είναι ο χρόνος που έχουμε για την ακρόαση. Τρία σκέλη ε, με παρουσιάσεις και μετά ένα γύρο ερωταπαντήσεων. Θα σας παρακαλέσω να είστε κάπως ε, σύντομοι στις παρεμβάσεις σας, δηλαδή ένα δίλεπτο ο καθένας για τις ερωταπαντήσεις και τώρα να ξεκινήσουμε την ακρόαση. Εάν ε, θέλετε θα δώσω το λόγο στο πρώτο τμήμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως κινητήριος δύναμη της Ευρώπης. Είναι όμως την πρώτη θέση. Ε, πρώτο τμήμα της ακρόασής μας να δώσω το λόγο στην πρώτη ομιλήτρια την κυρία Τζοάννα Ντρέικ. Τζοάννα ή Ιωάννα. Τζοάννα μάλιστα. Στη δική μου γλώσσα είναι Ιωάννα. Επίσης πολύ ωραίο όνομα. Ε, διευθύντρια και ειδική απεσταλμένη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στην DG ε, για τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα. Θα μας κάνετε μια παρουσίαση σε ένα δεκάλεπτο, εάν μπορείτε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπούζεκ Καλημέρα, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Ο κύριος Μπούζεκ ήδη είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκαθεν θεωρούσε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι προτεραιότητα για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που θα μας οδηγήσει σε περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Θα σας παρουσιάσω κάποια στατιστικά στοιχεία, ενδεχομένως τα γνωρίζετε ήδη, για να αποδείξω γιατί τα νούμερα δεν μας επιτρέπουν να πράξουμε διαφορετικά. 99 από τις 100 επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι μικρομεσαίες, 92 από αυτές είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δύο στους τρεις απασχολούμενους εργάζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 58 λεπτά σε κάθε ευρώ προστιθέμενης αξίας έρχεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει όμως και το μεγάλο αλλά. Στα περισσότερα κράτη-μέλη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν σε ένα οικονομικό περιβάλλον που υψώνει μεγάλες προκλήσεις μπροστά τους. Η ανάκαμψη ενδεχομένως υπάρχει, αλλά είναι ακόμα πολύ αδύναμη, μερική, τμήματική και δεν τους επιτρέπει να χαράξουν μια πορεία με δυναμισμό. Παρόλο που η αξία τους και ο αριθμός τους είναι πάνω από τα επίπεδα που υπήρχαν πριν από την κρίση, ωστόσο απασχολούν λιγότερους υπαλλήλους από ότι το 2008. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει δράση να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε την ομοθετική πράξη ε, για τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, Small Business Act, υιοθετήθηκε το 2008, αναθεωρήθηκε το 2011, είναι το βασικό εργαλείο ε, πολιτικής. πρέπει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε έτσι ώστε να έχουμε το βέλτιστο επιχειρηματικό περιβάλλον και να έχουμε σωστή χάραξη πολιτικής και σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να συνεχίσουμε ε, με αυτόν τον τρόπο ε, με τα επόμενα προγράμματα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλό θα είναι όμως να σας παρουσιάσω σύντομα τα επιτεύγματά μας αλλά και τις προκλήσεις που συνεχίσουν να υψώνονται μπροστά μας. Αρχικά μιλάω για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στην καινοτομία. Και εδώ πρέπει να πω το μεγάλο ευχαριστώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί εσείς είσαστε ο, κοινο, ο κινητήριος μοχλός πίσω από την αλλαγή παραδείγματος. Ε, την οποία ε, προσπαθήσαμε, την οποία καταφέραμε <clears throat> έτσι ώστε να στηρίξουμε την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντες 2020. Έχουμε ένα νέο εργαλείο, το εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στήριξη τριών δις για αυτές που έχουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και με προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, από τη βάση προς την κορυφή της πυραμίδας. Είναι σαφέστατο ότι πηγαίνουμε Προ τη σωστή κατεύθυνση γιατί το, αυτό το δείχνουν τα αποτελέσματα και σας τα παρουσιάζω ευθύ αμέσω, Μετά τον πρώτο γύρο αξιολόγηση και επιλογής των προτάσεων, το 70% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ε, θα τύχουν στήριξη στην πρότασή τους είναι για πρώτη φορά δικαιούχοι του προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη. Η ανανέωση δηλαδή της προσέγγισης μας μας έκανε να έχουμε πρόσβαση σε νέους ετούντε, σε νέους δικαιούχου. Και αξίζει να σημειωθεί το ότι το 1 τρίτο των επιχειρήσεων που στηρίζονται είναι νέες επιχειρήσεις, τριών ή πέντε ετών και θέλουμε να τις αποκαλούμε σταθεροποιημένες ε, startup, σταθεροποιημένες νεοσύσταθήσεις επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει ένα σημαντικό όραμα, έχουν χαράξει ένα όραμα, θέλουν να προχωρήσουν, θέλουν να αναπτυχθούν και ζητούν τον κατάλληλο μοχλό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτά τα δύο περιστατικά που μόλις σας ανέφερα, γιατί ερχόμαστε εμείς και προσφέρουμε αυτό το μοχλό εκτείναξης αν θέλετε. Πρέπει αυτοί οι προσανατολισμοί να γίνονται αντιληπτοί παντού και να προσελκύουμε τους πιο καινοτόμους επιχειρηματίες. Υπάρχει και το πρόγραμμα COSME με προϋπολογισμό 1,4 δις για τα χρηματοδοτικά ε, μέσα. Στοχεύει το πρόγραμμα COSME να βοηθήσει 330.000 ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι μάλλον ένα όριο που σίγουρα θα ξεπεράσουμε. Γιατί και με το προηγούμενο πρόγραμμα, το πρόγραμμα SIP, ε, βοηθήσαμε 360.000 ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και υπάρχουν κονδύλια τα οποία πρέπει να δαπανηθούν. Ωστόσο έχουμε ε, το στόχο, τον κατώτερο στόχο να βοηθήσουμε 330.000 ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις βάσει του προγράμματος COSME μέχρι το τέλος του. Και θέλουμε να κινητοποιήσουμε 21 δις χρηματοδότησης με μορφή δανεισμού και 3 δις χρηματοδότησης με τη μορφή επιχειρηματικών κεφαλαίων βάσει συμπράξεων. Και έχουμε θετήσει και το σχέδιο το επενδυτικό των 300 15 δις ευρώ που έχει ανακοινωθεί την περασμένη εβδομάδα έγινε αυτό από τον πρόεδρο ε, Γιούνκερ. Σημαντικό μέρος του επενδυτικού σχεδίου είναι η σύσταση ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις στρατηγικές επενδύσεις. Ήδη έχουμε βρει και το νέο όνομα του Ταμείου, το ΕΦΣΙ. Το Ταμείο λοιπόν θα χρηματοδοτήσει στρατηγικά projects σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ευρυζωνικές συνδέσεις, σε ενέργεια, σε μεταφορές, εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία κτλ και στόχος είναι να δοθεί νέα όθηση στην πραγματική οικονομία. Το 1 τέταρτο των πόρων θα αξιοποιηθεί για ε, τη χρηματοδότηση κινδύνου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και για τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και έτσι θα έχουμε επενδύσεις περίπου 75 δις ε, ευρώ επενδύσεων. 1 προς 13 θα είναι ο λόγος της μόχλευσης. Και αυτό θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις ελλείψεις κεφαλαίου. Θα έχουν υψηλότερα ποσά ίδιων κεφαλαίων, θα έχουν επιπρόσθετες εγγυήσεις για την ε, τιτλοποίηση υψηλής ποιότητας των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι αυτός ο αποτελεσματικός ε, τρόπος για να ενισχύσουμε τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη. Να σας πω τώρα για τη βιομηχανική πολιτική και τα clusters. Πρέπει να έχουμε μια ισχυρή βιομηχανική βάση με υψηλές ε, επιδόσεις στην εσωτερική αγορά έτσι ώστε το βάρος της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της Ένωσης να ξαναέρθει στο 20% μέχρι το 2020. Αυτό είναι κάτι που έχει δηλώσει ο πρόεδρος Γιούνκερ στο, ε, στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη νέα θητεία της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χαίρομαι διότι τα κράτη-μέλη στηρίζουν τις βασικές γραμμές αυτής της βιομηχανικής πολιτικής. Για παράδειγμα, η πολιτική αυτή τονίζει το πόσο δυναμικό έχουν τα κλάστερ για να έχουμε ευνοϊκά οικοσυστήματα για την καινοτομία, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν ανάγκες και θα πρέπει να να, ε, να καλυφθούν. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να παρουσιάσει το 2016 μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα κλάστερ, για τις συστάδες, για τις συμπράξεις, για την ανάπτυξη και έτσι θα έχουμε περισσότερη διατομεακή καινοτομία μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και διαπεριφερειακή συνεργασία. Και αυτό είναι σημαντικό για να ενισχυθεί η ανάπτυξη πρέπει να έχουμε ένα κανονιστικό περιβάλλον πιο ισορροπημένο, κανονιστικές διατάξεις που να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τους τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να μοιράζεται καλύτερα το βάρος ε, συμμόρφωσης στους νέους κανονισμούς και στις νέες διατάξεις. Αυτό σημαίνει μειώνω το διοικητικό ή γραφειοκρατικό άχθος. Και Πρέπει να σας πω ότι ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς στο, στην ομιλία που έβγαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια στις 24 Νοεμβρίου είπε ότι πρέπει να προωθήσουμε κανονισμούς και διατάξεις που ε, καταρρύπτουν τα εμπόδια προς την ανάπτυξη. Πρέπει να επιτρέψουμε σε νέες ευκαιρίες να αναδυθούν, να είναι η ανάπτυξη κοινωνικός και περιβαλλοντικός αϊφόρα. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε γιατί ξεκινούμε από μια στέρεα βάση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι στον πυρήνα του ε, προγράμματος ε, για την κανονιστική ε, επάρκεια και τις σωστές νομοθετικές επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το πρόγραμμα REFIT, έτσι ώστε να έχει fitness η νομοθεσία, να είναι η κατάλληλη, να είναι η ταιριάζει. Και πρέπει να κάνουμε και τα επόμενα βήματα έτσι ώστε να έχουμε πραγματικά ωφέλη για όλους τους επιχειρηματίες. Για παράδειγμα, πρέπει να είναι δυνατόν να ξεκινήσει κανείς, να ιδρύσει κανείς μια εταιρεία μέσα σε τρεις μέρες και με μέγιστο κόστος τα 100 ευρώ σε όλα τα κρατημέλη. Να μπορεί να πάρει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις μέχρι ε, μέσα σε ένα μήνα. Και μάλιστα αυτό είναι δύσκολο να γίνει, δυστυχώς. Η πρόκληση λοιπόν που υψώνεται μπροστά μας και αυτό που προτείνουμε είναι αυτά να γίνονται μέσα σε ένα μήνα. Πρέπει από εκεί και πέρα να καταρριφθούν αυτά τα εμπόδια και ε, η αίτηση για το SME test, για το τεστ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να είναι υποχρεωτική ή κάποιο αντίστοιχο σύστημα να είναι υποχρεωτικό σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γνωρίζουμε να γνωρίσουν όλοι ε, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος του κανονισμού αυτού στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πρέπει και να φροντίσουμε τις επιχειρήσεις που πτωχεύουν να έχουν τη δυνατότητα να ξαναξεκινήσουν, να τους δοθεί μια νέα, μια δεύτερη ευκαιρία. Και θα πρέπει να υπάρχει ένα, ένας χρόνος απαλλαγής, ε, μέγιστος χρόνος τριών ετών για τους επιχειρηματίες. Mm. Έρχομαι τώρα στην πρόσβαση στις αγορές. Ζούμε σε μια τεράστια αγορά, τη μεγαλύτερη αν θέλετε του κόσμου και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούν ότι όντως αυτό πρέπει να είναι το γήπεδο στο οποίο πρέπει και να μπορούν να παίξουν μπάλα και μάλιστα χωρίς εμπόδια και καλώς. Έχουμε το δίκτυο ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ΕΕΝΗ, ε, αυτό διαδραματίζει ένα σημαντικό, ένα καθοριστικό ρόλο έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που δεν έχουν απαραίτητες πληροφορίες για τη νέα αγορά τη νέα ενιαία αγορά να μπορούν εκεί να τις βρουν συγκεντρωμένες γιατί δεν υπάρχει χρόνος ή δεν υπάρχει δυνατότητα να επισκέπτονται διαφορετικές ιστοσελίδες και να αναζητούν την πληροφόρηση σε διαφορετικές ε, πηγές. Και έτσι πρέπει να τους διευκολύνουμε να έχουν και να μπορούν να αδράξουν αυτές τις επιχειρηματικές ευκαιρίες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέρα από αυτές. Πρέπει λοιπόν να επιδιώξουμε να συνεχίσουμε αυτές τις ε, προσπάθειες όσο περισσότερο μπορούμε. Γιατί οι εξαγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι και οι πιο ανταγωνιστικές, γιατί είναι οι πιο παραγωγικές, οι πιο καινοτόμες και διαθέτουν ε, προσωπικό με τις περισσότερες και καλύτερες δεξιότητες και προσόντα. Η γενική μας διεύθυνση δεν θα είναι πια γενική διεύθυνση επιχειρήσεων ή επιχειρηματικότητας, θα αλλάξει όνομα, θα είναι DG Grow, θα είναι γενική διεύθυνση για την ανάπτυξη. Θα έχει καινούργια ονομασία από τον Ιανουάριο της επόμενης χρονιάς. Και το κάνουμε αυτό διότι ε, θεωρούμε ότι πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο για ε, επιχειρηματικότητα, για καινοτομία, για έξυπνες ιδέες να βοηθήσουμε έτσι ώστε να υπάρξει συνεργασία και συνέργεια για να γίνουν όλα αυτά στην πράξη. Κύριε Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει μια σταθερή, μια στέρεα πολιτική έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συνεχίζουν να βρίσκονται πίσω από την ανάπτυξη και την απασχόληση, να βρίσκονται στο τιμόνι, να συνεχίσουμε να τους επιτρέπουμε να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα από όλα. Και πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε ε, το Small Business Act, το βασικό νομοθετικό εργαλείο που έχουμε αυτή τη στιγμή, και το κάνουμε, το αναθεωρούμε, το επανεξετάζουμε για να τις βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο. Να σας υπενθυμίσω ότι μια δημόσια διαβούλευση, αυτή που εκτελήσεται αυτή τη στιγμή, θα ολοκληρωθεί στα μέσα του Δεκεμβρίου για την αναθεώρηση αυτού του νομοθετήματος και το νέο, η νέα νομοθετική πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις θα παρουσιαστεί ε, στο πρώτο εξάμεινο του 2015 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκαθεν στηριζόμασταν στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε έτσι ώστε αυτό το νομοθετικό μέσο να δίνει προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μας οδηγήσουν σε περισσότερη ευημερία και ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Τζέικ για την παρουσίασή σας για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Πατρίσια Κάλλαν. Τώρα μπαίνουμε πραγματικά στο χώρο των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διότι εσείς εκπροσωπείτε την Ένωση Μικρών Επιχειρήσεων της Ιρλανδίας. Οπότε, έχετε γνώση της θέσης πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας σας και πολλών άλλων χωρών, καθώς έχετε πολλές επαφές και με άλλες ενώσεις. Έχετε το λόγο, κυρία μου. Καλημέρα σε όλους, πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την Γιακόλη που με έφερε ε, και με προσκάλεσε να μιλήσω εδώ σήμερα το πρωί. Είναι μεγάλη μου χαρά να μπορώ να σας μιλήσω για τις δικές μας εμπειρίες από τα μέλη της Ένωσής μας στην Ιρλανδία και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην παρουσίασή μου σήμερα το πρωί ήθελα να σα δώσω κάποιε λεπτομέρειε για τι μικρέ επιχειρήσει στην Ιρλανδία και πώ πάνε εκεί τα πράγματα και μετά θα δούμε τι γίνεται με τα μέλη τη Ένωσή μα, τι μα λένε οι επιχειρήσει που δουλεύουν καθημερινά στην πράξη, στην αγορά, γιατί ε, ήταν ένα θέμα να επιβιώσουν από την κρίση οι εταιρείε αυτέ και να περάσουν πάλι σε ε, τροχιά ανάπτυξη. Επίση, θέλουμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε εσεί οι Ευρωβουλευτέ, τι προσπάθειέ του, να του στηρίξετε στι προσπάθειέ του, για να ε, περάσουν πάλι σε τροχιά ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσει εργασία. Ω προ τη δική μου την Ένωση, υπάρχουμε για να ακουστεί η φωνή των μικρών εταιριών στην Ιρλανδία και διεθνώς με περίπου 8.000 εταιρείε σε όλους τους τομείς, σε όλη τη χώρα στην Ιρλανδία, δίνοντάς τους συμβουλές για το πώς να λειτουργήσουν καλύτερα, αλλά και για άλλα πράγματα όπως τη συμμόρφωση με την νομοθεσία ή τους νόμους ε, για την εργασία και έχουμε ένα πολύ καλό δίκτυο για να μπορέσουν οι εταιρείε να συνεργαστούν καλύτερα μεταξύ τους και πολλές φορές να εκπροσωπηθούν και δημοσίως εφόσον χρειαστεί για βασικά ζητήματα. Ω προ την Ελληνδία, λοιπόν, ο ορισμό που χρησιμοποιώ για τι μικρέ επιχειρήσει είναι ε, μια εταιρεία που απασχολεί λιγότερου από 50 εργαζομένου. Στην Ιρλανδία και στην Ευρώπη, λοιπόν, γενικώ, ο όρο ε, μικρομεσαία επιχείρηση σημαίνει κάτω από 250 εργαζομένου. Όμω στην Ιρλανδία λέμε ότι οι μικρομεσαίε ε, διαφε... διαφέρουν. Διαφέρουν διότι έτσι κι αλλιώς η χώρα είναι μικρότερη. Όμως σε κάθε χώρα ε, περίπου τα στατιστικά στοιχεία είναι, δηλαδή οι αυτοαπασχολούμενοι, αυτοί που απασχολούν το πολύ τρεις ανθρώπους, ε, είναι ε, το πιο σύνηθες και οι περισσότεροι είναι αυτοί που κινούν την εγχώρα οικονομία κάθε χώρας, δεν εξάγουν και τους δημιουργεί προβλήματα το γεγονός ότι όλη η έμφαση δίνεται στις νέες τεχνολογίες, στις ε, νεοφυείς που χρησιμοποιούν καινοτόμε μεθόδους και εξάγουν. Εδώ χρειάζονται και αυτή τη στήριξη, διότι επιχειρήσεις χρειαζόμαστε σε κάθε κλάδο και τομέα της οικονομίας. Βεβαίως, αν μπορέσουν και αυτές οι εταιρείε να ε, αναπτυχθούν και να εξάγουν, θα είναι πάρα πολύ καλό. Όμως ήδη η δουλειά που κάνουν με έναν, δύο, δέκα, είκοσι εργαζομένους είναι εντυπωσιακή. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ω προ την αίσθηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπω είπε και η Τζοάννα, νομίζω ότι τα πράγματα ε, ε, περνάνε σε μια φάση σταθερότητα. Έτσι το αντιλαμβάνεται το κοινό. Ότι μπορεί να περάσουμε πάλι σε ανάπτυξη. Οι αριθμοί αυτοί, που δεν είναι ακόμα πάρα πολύ αισιόδοξοι, τουλάχιστον δείχνουν 50% των μελών μα να θεωρούν ότι οι δουλειέ του πάνε καλά ή πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Βλέπουν τεράστια ε, εντύπωση σχέση, ε, τεράστια βελτίωση μάλλον, σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από 12 μήνε. Ω προ τι αλλαγέ τη εκτιμήσει μα στην ε, Ιρλανδία, στις προβλέψεις μας, βλέπουμε να υπάρχει ένα εφικτό 3-4% ποσοστό ανάπτυξης για τα επόμενα 3-4 χρόνια σε σχέση με την κατάσταση ε, από την οποία βγήκαμε, δηλαδή το πρόγραμμα διάσωσης της Τρόικας. Ε, ο λόγος που το βλέπουμε αυτό είναι ότι πείσαμε την κυβέρνηση και χαίρομαι που και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, σε μια φάση δηλαδή που αναγνωρίζουμε ότι η λιτότητα δεν ε, είναι κάτι που πρέπει να διαρκέσει, διότι εκείνη τη στιγμή που χρησιμοποιήθηκε ίσως ήταν ε, απαραίτητη, όμως αν θέλει κανείς να ξεφύγει από δυσχερείς οικονομικές καταστάσεις πρέπει να λάβει μια όθηση. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που να ευνοεί τις επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις να λειτουργούν, να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και αυτές να συνεισφέρουν στην φορολογία. Φορολογία που μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι κυβερνήσεις για να, αναδια... να... να διανύμουν τα έσοδά και να καλύψουν κοινωνικές ανάγκες. Αυτό πρέπει να έχουμε λοιπόν στο μυαλό ε, κατά όταν συζητούμε τις πολιτικές μας επιλογές. Είναι ένα βασικό μήνυμα ότι πρέπει να επενδύσουμε για να λάβουμε και το ε, κέρδος, το όφελος από τις επενδύσεις μας. Ως προς τα διδάγματα από την κρίση νομίζω ότι αυτά είναι σημαντικά για τις εταιρείε όλης της Ευρώπης και κάτι που θέλω να μοιραστώ και μαζί σας σήμερα το πρωί είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν ξέρουν τι συμβαίνει εδώ. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει ούτε καν στα εθνικά κοινοβούλια. Ε, ουσιαστικά κοιτάζουν ε, την καθημερινή τους δουλειά και θέλουν να μπορούν να το κάνουν αυτό χωρίς να τις εμποδίζουν οι κυβερνήσεις. Ε, εάν γίνεται μάλιστα να διευκολύνουν και να μπορούν να επιλύουν με θετικό τρόπο τα πολιτικά ζητήματα. Αλλά δεν ξέρουν τις λεπτομέρειες το τι αποφασίζεται εδώ ή από τις κυβερνήσεις ξέρουν απλώς εάν κάτι τους βολεύει ή όχι, αν είναι λάθος ή σωστό. Αυτό λοιπόν που, κάνουν επιχειρήσεις, ε, που έκαναν οι επιχειρήσεις στην κρίση είναι ότι πήραν τα πράγματα στα χέρια τους, πήραν γρήγορα πολύ κέρυες αποφάσεις όπως απολύσεις, ε, περικοπές τους μισθούς, ε, τη διατήρηση του βασικού πελατολογίου και ε, την διατήρηση της βασικής παραγωγής. Αυτό για να ελέγξουν ε, το κόστος. Είδαμε τεράστια, τεράστια κέρδη στην ανταγωνιστικότητα στην Ιρλανδία και νομίζω και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να δούμε τι κόστος επιβάλλουν οι κυβερνήσεις για να προσπαθήσουμε αυτό το κόστος να περιορίσουμε. Οι κυβερνήσεις πολύ συχνά ε, αποφασίζουν τις τιμές σε χώρους όπως η ενέργεια, η φορολογία, η άλλα εμπορικά ε, θέματα. Στην ε, ε περίπτωση του συστήματος υγείας λόγω χάρη, της, του εκπαιδευτικού συστήματος, εκεί θέλουμε να μην υπάρξει μια πολλαπλασιαστική εκτός ελέγχου αύξηση του κόστους. Πάντως, η χρηματοδότηση είναι το βασικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη όλα τα νέα ε, δημοσιονομικά και χρηματοδοτικά εργαλεία ε, είναι ευπρόσδεκτα και η χρηματοδότηση από το κόσμο. Ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα εκ μέρου του Κοινοβουλίου. Αυτό που χρειάζονται όμω οι μικρέ εταιρείε στην Ιρλανδία και πιστεύω και σε όλη την Ευρώπη, ε, το χρειάζονται και του απογοήτευσε ότι επί τη ουσία ε, ο μηχανισμός, ε, οι μηχανισμοί λειτουργούν μέσω των υπαρχόντων ε, ε μεσαζόντων που είναι ήδη γνωστοί. Δηλαδή στην τράπεζα, είτε το, η χρηματοδότηση προέρχεται από το κόσμο είτε από αλλού, πρέπει να πάει κανείς στην τράπεζα, είτε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είτε μια εμπορική τράπεζα, πρέπει να πάει κανείς στο ίδιο άτομο που ήξερε και πριν. το άτομο αυτό είναι που θα λάβει την απόφαση εάν θα στηρίξει εσένα και την επιχείρησή σου. η εμπιστοσύνη λοιπόν και το επίπεδο εμπιστοσύνη πολιτικό πολιτών στου τράπεζέ μας, που δεν καταλαβαίνουν την περίπλοκη λειτουργία κάποιων εταιριών, που δεν είναι έτοιμε να υποστηρίξουν αναγκαστικά πρόσωπα ή ε, λειτουργία επιχειρήσεων, αλλά να ζητούν εγγυήσει ε, αντί, αντίτιμα και ανταλλάγματα για να χρηματοδοτήσουν, αυτό δημιουργεί πρόβλημα στις ε, εταιρείε. Λόγω χάρη στα Ιρλανδικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι πολίτες ξέρουν ότι υπάρχουν ε, στατιστικά στοιχεία, ε, αριθμητικά στοιχεία που αναγκάζουν να πάνε τους διάφορους διαμεσολαβητές για να βρουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται για την αγορά. Θα περάσω σε περισσότερε λεπτομέρειε γι' αυτό και στη συνέχεια, αλλά αυτό είναι το βασικό θεμελιώδε πρόβλημα. Το πώ εκτιμά η τράπεζα τον κίνδυνο λειτουργία τη κάθε ε, εταιρεία. Επίση, πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στο ανθρώπινο κεφάλαιο, του ανθρώπινου πόρου. Γι' αυτό, στο πλαίσιο τη συζήτηση που κάνουμε για, τις, ε, για το Small Business Act στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου, του μάνατζερ. Είδαμε ότι το 50% οι μισέ μικρέ εταιρείε συνήθω αποτεχάνουν την πρώτη πενταετία. Όμω θα μπορούσαμε να μειώσουμε στο μισό αυτό το ποσοστό αν είχαμε επενδύσει στο, στη διεύθυνση τη εταιρεία. Και υπάρχουν διεθνεί δείκτε γι' αυτό. Η χρηματοδότηση για την κατάρτιση συνήθω τρέφεται προ του ανέργου. Δεν ε, καλύπτουμε αυτού που έχουν δεξιότητε, αλλά αυτού που δεν έχουν. Θα έπρεπε όμω να επενδύσουμε επενδύσουμε περισσότερο στους επιχειρηματίες ενδεχομένως, τους μάνατζερ και αυτούς που ήδη δουλεύουν. Όπως με τις ε, χρηματαγορές, το είδαμε και στην κρίση, αυτοί που ευνοήθηκαν ήταν οι τολμηροί, αυτοί που πήραν αποφάσεις, που στην αγορά κινήθηκαν γρήγορα και πέτυχαν κέρδο. Έτσι μπορεί να λειτουργήσει μια νεοσύστατη εταιρεία με καινοτομία για την καινοτομία, όπω συνήθω οι περισσότεροι άνθρωποι ε, το ταυτίζουν με τι ε, τεχνολογίε αιχμή. Δεν είναι όμω μόνο έτσι. Μια μικρή εταιρεία λιανική, ένα μικρό ξενοδοχείο, ένα μικρό εστιατόριο, ε, μια μικρή μεταποιητική εταιρεία. Κάθε επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει τι επιδόσει τη εφόσον οι άνθρωποι βελτιώσουν λόγω χάρη το customer service που παρέχουν, τι υπηρεσίε προ τον πελάτη, την εξυπηρέτηση πελατών. Έχουμε ένα πρόγραμμα, το λεγόμενο Innovation Voucher, τα δελτία για την καινοτομία που επιτρέπουν στις εταιρείες να ζητήσουν βοήθεια για να προωθήσουν τις, ε, τη λειτουργία τους. Ω προ τι προτεραιότητέ μα τώρα, καθώ προχωρούμε, ζητήσαμε από μια σειρά από εταιρείε να μα πούν ποιο από αυτού του πέντε παράγοντε θα μπορούσε περισσότερο να συμβάλλει στην ε, ανάπτυξή του. Το ενδιαφέρον είναι ότι περίπου τα ίδια ποσοστά πήραν οι πέντε αυτέ επιλογέ. Δηλαδή, ε, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ότι το 11% της ανεργίας στην Ιρλανδία είναι ένα μεγάλο θέμα, παρόλο που το ποσοστό είναι μεγάλο στην, ε, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρόλα αυτά έχουμε έλλειμμα δεξιοτήτων. Δεν μπορούμε δηλαδή να καλύψουμε τις ανάγκες του τομέα της τεχνολογίας, λόγω χάρη. Πολλέ φορέ χρειάζεται να φέρουμε μετανάστε λόγω χάρη στον τομέα τη υγεία. Αυτό θα πρέπει να το ισορροπήσουμε καλύτερα. Όμω, στη δεύτερη θέση, πολλοί ανησυχούν και για τι προοπτικέ ανάπτυξη εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε τυχεροί που στην Ιρλανδία έχουμε πολλέ συναλλαγέ με το Ηνωμένο Βασίλειο και τι Πολιτείε, Όμω, θα θέλαμε, θα θέλαμε και μια σταθερότερη ανάπτυξη από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, εσωτερικά θα πρέπει να έχουμε ένα περιβάλλον φορολογικό πιο ευνοϊκό προ τι επιχειρήσει ως προς το τι αναζητούν ε, οι άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν, ε, ως προς τα προγράμματα θα θέλαμε επενδύσεις όπως ε, τις εταιρείε που θέλουν να αναπτύξουν την, την, το σήμα τους ή την, το ανθρώπινο δυναμικό ως προς τις προτεραιότητές μας είναι παρόμοιες με τι εταιρείε οποιοδήποτε άλλο ένωση ενό άλλου κράτου μέλου. Πρέπει να δούμε πώ θα στηρίξουμε την εσωτερική ζήτηση, την εγχώρια ζήτηση, πώ θα στηρίξουμε τι εγχώριε εταιρείε, τη δημιουργία θέσεων απασχόληση εσωτερικώ και πώ θα μείνουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει στην καρδιά τη ε, χάραξη νομοθεσία. Διότι δεν ξέρω αν οι περισσότεροι όταν ε, λαμβάνουμε θετικέ αποφάσει σκέφτονται πρώτα τι ε, ανάγκε των μικρών. Θα πρέπει λοιπόν να μειωθεί και το κόστο τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα και οι δημόσιε προμήθειε, οι διαγωνισμοί. Τα κονδύλια στη Γερμανία έχουν ε, ένα πολύ καλό τρόπο να στηρίζουν τις ε, εταιρείε μέσω των ε, δημόσιων διαγωνισμών, έτσι όπως προβλέπεται το σύστημα. Πρέπει να ισχύει και στην Ιρλανδία, παρόλο που κανόνες υπάρχουν, να επιβάλλονται κανόνες ή να αλλάξουν, ώστε οι μικρές εταιρείε πραγματικά να μπορούν να συμβάλλουν. Και να έρθω και πάλι στους νόμους εργασίας και απασχόλησης. Πολλές αποφάσεις νομοθετικές λαμβάνονται και εδώ. Εάν θέλετε να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας, διευκολύνεται τις εταιρείε να προσλάβουν κόσμο. Εάν έχει κανείς μια εταιρεία και πρέπει να ξέρει απ' 40 νομοθετήματα, προβλήματα, ασχέτω με το απόσχολη, αποσχολεί, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να ξέρετε ίδια με κάποιον που έχει 5.000 εργαζόμενου. Ε, άρα, επί τη αρχή, ξέρω ότι έχει τελειώσει ο χρόνο μου, οπότε θα τη δείξω κατευθείαν στην τελευταία μου διαφάνεια. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει. Να, νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ε, τις πολύ μικρές εταιρείε. Δηλαδή όχι γενικά μικρομεσαίες. Οι μεσαίες επιχειρήσεις έχουν πολύ διαφορετικές ανάγκες από τις μικρές και τις πάρα πολύ μικρές. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε γιατί η απασχόληση από αυτές θα προέλθει. και όπως το είπε και Τζοάννα προηγουμένως, τα βλέπετε και στη διαφάνεια σε ανακεφαλαίωση, αλλά πραγματικά πρέπει να μειωθεί το γραφειοκρατικό άκθο, να βελτιωθεί η πρόσβαση στι αγορέ, να τονωθεί η επιχειρηματικότητα. Με χαρά να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε, αλλά ελπίζω ότι αυτέ οι πληροφορίε που σα έδωσα από τι εταιρείε που είναι μέλη τη Ενωσή μα ήταν χρήσιμε σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι ευκαιρίε για πράσινη ανάπτυξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο κύριος Ντεμπάκερ, ο εισηγητής μας, θα πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τους δύο μιλητές για την έκκληση, την παθιασμένη που μας απέφθηναν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι έχουμε ανθρώπους ε, μαζί μας ε, που προασπίζουν τα σημεία τα οποία και εσείς παρουσιάσατε. Να ξεκινήσω από την αγανάκτηση της τελευταίας ομιλήτριας όταν αναφερθήκατε στα διάφορα φορολογικά καθεστώτα, στα, στις διάφορες εργασιακές νομοθεσίες που δυσκολεύουν όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην υποτιθέμενη ενιαία αγορά. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει μια συζήτηση και σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Μια συγκεκριμένη ερώτηση έχω να κάνω και στους δύο σας γνωρίζουμε ότι ιδιαίτερα στο θέμα του περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μεγάλη νομοθεσία. Καταρτίζουμε μεγάλη νομοθεσία. Προσπαθούμε η νομοθεσία αυτή να είναι το όσο πιο αποδεκτή γίνεται για τις επιχειρήσεις, αλλά πρέπει να θέτουμε και στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο παράλληλα. Έχουμε συζητήσει θέματα καλύτερης ρυθμίσης, καλύτερης νομοθεσίας, εφιέστερη νομοθεσία. Τώρα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει θέσει ως στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ίσως θα πρέπει να υπάρχει και μείωση της νομοθεσίας, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση υπάρχει και η συζήτηση για το κατά πόσο θα μπορούσαν και θα έπρεπε να εξαιρούνται από κάποιες νομοθεσίες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε στην περίπτωση που δεν θα υπάρχει αυτή η παρέκκληση ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις ε, σύνθετες συνθήκες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ροϊμπίχ είναι ο σκιώδης συζητητή μα και επικεφαλής του ΣΤΟΑ που από πλευρά κοινοτομία θα μπορούσε επίση να υποστηρίξει τι ε, μικρομεσαίε επιχειρήσει μα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρωτοβουλία σα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να φροντίσουμε στην Ευρώπη να παράγουμε προϊόντα και να παρέχουμε υπηρεσίες οι οποίες να είναι επιθυμητέ σε παγκόσμιο επίπεδο και προς αυτή την κατεύθυνση χρειαζόμαστε και την υποστήριξη των απαραίτητων υποδομών. Στην ψηφιακή αγορά προσπαθούμε να την οργανώσουμε με τέτοιο τρόπο, όπως και την ενεργειακή αγορά άλλωστε, καθώς και το θέμα της ε, στρατηγικής για την ενιαία αγορά. Θα πρέπει όλα αυτά να έχουν σκοπό την ανταγωνιστικότητα. Και το δημόσιο σκέλος ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ε, τα μοντέλα ιδιωτικών και δημόσιων σε, συμπράξεων θα πρέπει να προωθηθεί η στρατηγική αυτή. Θα πρέπει τα έσοδα να είναι πιο υψηλά από τις δαπάνες της επιχειρήσεις. Αυτό πλέον σήμερα ξέρετε δεν είναι δεδομένο, αλλά στις σπουδές μου, τις πενταετής σπουδέ μου για θέματα οικονομικά, έμαθα ότι μόνο όταν υπάρχει κέρδος μπορούμε να μιλάμε για κεφάλαιο κινδύνου. Μόνο αν υπάρχει κεφάλαιο κινδύνου μπορεί να πάρει κανείς πιστώσεις και μόνο αν υπάρχουν πιστώσεις μπορεί κανείς να έχει εγγυήσει για τις συναλλαγές, για τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν de facto αυτό το θέμα να το πραγματευτούμε. Αυτό είναι το θέμα σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα. Αυτό το κεφάλαιο κινδύνου λοιπόν στις επιχειρήσεις θα πρέπει να υπάρχει, να είναι στεναρό. Ξέρουμε ότι η φορολογία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, είναι πολύ υψηλή. 80% των φόρων που λαμβάνουμε στην Ευρώπη προέρχονται από τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και βλέπουμε ότι οι διεθνοί όμιλοι πληρώνουν μόνο 4%. Νομίζω ότι υπάρχει λοιπόν μια αναλογία, μια σοβαρή αναλογία. Θα πρέπει να φροντίσουμε οι μικρομεσαίες επιχειρήσει να πληρώνουν εξίσου χαμηλού φόρου όπω οι μεγάλοι όμιλοι. Μόνο τότε θα μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικές και έτσι να αυξηθούν, να αναπτυχθούν με επιτυχία. Αυτό είναι το έργο της νέας Γενικής Διεύθυνσης. Να υποβοηθήσει την ανάπτυξη, να αναπτυχθεί το κεφάλαιο κινδύνου και με το κεφάλαιο κινδύνου να υπάρχει μια κινητήρια δύναμη, ένας μοχλός για να, λάβουν, να λαμβάνουν πιστώσεις, γιατί χωρίς ίδιο κεφάλαιο δεν προβλέπεται η δυνατότητα δανεισμού. Αυτό το προβλέπει η Βασιλεία 3 και έτσι σε τελική ανάλυση έχουμε αυτούς τους ε, κρυφούς πρωταθλητές ε, ε, μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα, οι οποίες είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό, αλλά έχουν ως στόχο να κατακτήσουν τη διεθνή αγορά. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες και αγοργά αναπτυσσόμενες εταιρείε προκειμένου να βελτιώσουμε τους όρους λειτουργίας τους και σε ό,τι αφορά ε, τη συνθήκη του ΠΟΕ που ελπίζουμε σύντομα να επικυρωθεί σε ό,τι αφορά τις ε, εμπορικές ε, διευκολύνσεις και φυσικά οι διμερείς σύμφωνίες που είναι πολύ σημαντικές ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για να υπάρχει επιτυχία σε διεθνές επίπεδο. Τελευταίο σημείο, η Γαλλία δημιούργησε 10 ε, αφορολόγητες ζώνες για επιχειρήσεις που μπορούν να ξεκινήσουν να συσταθούν χωρίς φορολογία προκειμένου να μπορέσουν να σχηματίσουν αυτό το κεφάλαιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Λεβαντόφσκι. Πριν από δύο έτη ήταν υπεύθυνο για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο για όλα τα χρήματα του ορίζοντα 2020 κόσμο, τα διευθυντικά ταμεία, πολλά χρήματα λοιπόν που κατέληγαν στα χέρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Πρέπει όντω να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό στην Ευρώπη και τα διάφορα ε, ελλείμματα που υπάρχουν. Αλλά ό,τι και να πούμε, Ακόμη και αν ο πολιτικό μα τόνο είναι ορθό, η κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη δεν είναι πολύ ικανοποιητική, ιδίω στην νότια, κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Όπου ουσιαστικά αυτοχρηματοδοτούνται οι επιχειρήσει και συνολικώ. Αυτό που δείχνει ότι οι νέε γενιέ αναλαμβάνουν κίνδυνο και μπορούν να αναλάβουν κίνδυνο είναι ότι οι νέε γενιέ μεταναστεύουν. Μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Το ίδιο ισχύει και για την Ιρλανδία. Έτσι, στην Ευρώπη έχουμε πολύ μετριοπαθή χρηματοδοτικά εργαλεία. Είμαστε πολύ μαζεμένοι για το ρυθμιστικό λοιπόν πλαίσιο. Αυτό που ήθελα να μου πείτε είναι για δύο από τα νομοθετήματα του ρυθμιστικού πλαισίου, κάτι που ανέφερε και ο κύριος Ρούμπικ. Ο κρίκος που απουσιάζει στην νομοθεσία μας για την απορρόφηση είναι αυτό που ονομάζουν ε, τα θεσμικά όργανα κεφάλαιο κινδύνου. Κάτι πρέπει να γίνει από νομοθετική άποψη και γι' αυτό και έπειτα για την ανάληψη κινδύνου. Είναι διαφορετικές, διαφορετική πρόσληψη της αποτυχίας στις διάφορες νοοτροπίες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η αποτυχία είναι μέρος της επιχειρηματικής δράσης. Αλλά ανάφεραν και δύο μιλήτριες ε, ε, το στοιχείο αυτό. Δηλαδή, την καταστροφή ας πούμε, την αποτυχία, πώς μπορεί κανείς να τη μετατρέψει σε ευφύη προσγείωση, σε μια ομαλή συνέχιση της προηγούμενης ζωής του και των δραστηριοτήτων του. Ευχαριστούμε κύριος Γκέρεκ. Από μια περιοχή άκρος βιομηχανική με πολλές μικρομεσαίες. Ευχαριστώ πρόεδρε μικρομεσαίε επιχειρήσει θα έπρεπε να, να χωριστούν σε δύο διαφορετικές κατηγορίε τι μεταποιητικέ και τι ε, εταιρείε που προσφέρουν υπηρεσίε. Αυτέ που προσφέρουν υπηρεσίε πιο εύκολα ενδρύονται και πιο δύσκολο είναι να υπάρξουν νεοσύστατε στον τομέα το μεταποιητικό, διότι ο εξοπλισμό κοστίζει περισσότερο, το κεφάλαιο για να ξεκινήσει κανεί είναι μεγαλύτερο και νομίζω ότι αυτή η διάκριση πρέπει να γίνει γιατί είναι σημαντική. Σήμερα Ο καθένα κάτι παράγει στον κόσμο. Όλοι θέλουν κάτι να κατασκευάσουν και να το πουλήσουν. Η αγορά ήδη φαίνεται κορεσμένη. Πώς λοιπόν να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να φτάσουν, να ανοίξουν δρόμο και να πάρουν μια θέση, να αποσπάσουν μια θέση σε μια τέτοια αγορά. Αν έχει κανείς μια μικρή ε, παραγωγή λόγου χάρη, αλλά εξαρτάται από μεγάλα δίκτυα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ιδάλλως είναι πολύ δύσκολη αρχή. Το κόσμο, το ΕΦΣΥ είναι σημαντικά προγράμματα και νομίζω ότι αυτά τα εφαλτήρια μπορούν να δώσουν ε, κάποια πρώτη στήριξη στις επιχειρήσεις. Όμως το νομοθετικό περιβάλλον και το πώς αντιλαμβανόμαστε τα θέματα αυτά και αναλόγως νομοθετούμε είναι πολύ σημαντικό. Τα θέματα λόγου χάρη της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν να κάνουν πολύ με την δράση των νεοσύστατων. Σε ό,τι αφορά τις ε, πολωνικές μικρομεσαίες λόγου χάρη, το δίπλωμα ευαισθητεχνίας που έχουν εγκρίνει 25 χώρες δυσχεραίνει τα πράγματα για τις μικρομεσαίες, διότι αν θέλει να επενδύσει μια εταιρεία, δεν ξέρει μήπως παραβεί κανένα νόμο πνευματικής ιδιοκτησίας ή όχι. Έπειτα υπάρχει και τεχνογνωσία για, το, για τα θέματα του εμπορίου προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα, ένα ακόμα μονοπόλιο εδώ νομίζω και όσο περισσότερα μονοπόλια υπάρξουν τόσο πιο δύσκολο είναι να ε, ιδρυθούν νέες εταιρείες στον τομέα των μεταποιητικών. Το εμπόριο, το εμπορικό απόρριτο είναι ένα από τα προβλήματα και αυτά θα πρέπει να δούμε με προσοχή. Κατά την άποψή μου πρέπει να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο περιβάλλον και σε επίπεδο τοπικών κυβερνήσεων και στα κρατημέλη που να ευνοεί, να ευνοεί την, ε, την δημιουργία τοπικής βιομηχανικής παραγωγής. Η βιομηχανία εφόσον δημιουργηθεί και σε εθνικό επίπεδο μπορεί να καλύψει τα κενά της αγοράς, όμως σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει εκεί να υπάρξει στήριξη. Το περιβάλλον εκεί να είναι ευνοϊκό πριν υπάρξει εξέλιξη. Συνάδελφοι, παρακαλώ να μείνουμε στο δίλεπτο. Ο σκιώδης εισηγητής από την ε, ο κύριος Λάνστορφ αλλά ε, και ο κύριος Σιλικιώτης ε, θα λάβει το λόγο γιατί θα αντικαταστήσει το σκιώδη συγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επειδή απουσιάζει ο σκιώδη συγητής ο κύριος Ραμστοφ ε, θα μιλήσω εγώ στη θέση του. θα ρωτήσω δηλαδή. Ε, ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τράκε και την κυρία Γκάλα για τις πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις τους. Όλοι συμφωνούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά και την κινητήρια δύναμη της οικονομίας μας Γι' αυτό είναι αδύρυτη ανάγκη να προωθηθούν πολιτικέ που στόχο έχουν να στηρίξουν τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Η ερώτησή μου απευθύνεται στην κυρία Ντράκε, η οποία θα ήθελα να μα πει εάν η Κομισιόν μελετά συγκεκριμένα μέτρα για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε εκείνε τι χώρε οι οποίε ε, επηρεάζονται περισσότερο από την οικονομική κρίση και αναφέρομαι κυρίως στις χώρες του Νότου, ε, στις οποίες εφαρμόζονται κατά την άποψή μα βάρβαρες μνημονιακές πολιτικές και βλέπουμε μικρομεσίες επιχειρήσεις κάθε μέρα η μια μετά την άλλη να οδηγούνται ε, στο κλείσιμο και να, να ενισχύουν έτσι να οδηγούν ε, πολλούς εργαζόμενους στην ανεργία. Τι είναι εκείνα τα μέτρα που πρέπει να παρθούν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από την δεσπέζουσα θέση που έχουν στην αγορά οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Και εδώ συμφωνώ με την κυρία Γκάλαν, εκείνε που χρειάζονται περισσότερη στήριξη είναι πολύ μικρέ επιχειρήσει, γιατί καμιά φορά όταν μιλούμε για μικρομεσαίε επιχειρήσει, ε, αναφερόμαστε και σε επιχειρήσει άλλε που έχουν τη δυνατότητα, ενώ πολλέ μικρέ επιχειρήσει δεν έχουν τα μέσα, δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε ε, χρηματοδοτικά εργαλεία. Το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω, κυρία Τράγκεν Αναφερθήκατε στο Ταμείο για Στρατηγικές επενδύσει, Μιλήσατε βέβαια για τα 75 δισεκατομμύρια. Γύρω που μπαίνει να ξεκαθαριστεί είναι η συμβολή ιδιαίτερα της, ε, ε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2012 ξεκίνησε μια συζήτηση για τις κρατικές ενισχύσεις και πρέπει να το γνωρίζουμε χωρίς να συμμετέχει το κράτος, χωρίς να συμμετέχει και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι δίνεται να ε, κάτω από το βάρο της κρίσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τρέσα Γκρίφιν, η οποία είναι μεγάλη υποστηρίκτρια της κοινοτομίας, αν θυμάμαι καλά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τζοάννα, μιλήσατε για την στρατηγική κλάστερ για την ανάπτυξη. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι αυτά που μας περιέγραψε η Πατρίσια και τα διδάγματα θα ε, εισέλθουν στη νέα στρατηγική για την ανάπτυξη οι ανάγκες των μικρομετουσαίων επιχειρήσεων γιατί όπως ε, ανέφερε και η Πατρίσια υπάρχει ομαδοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι οικονομικοί διαμεσολαβετές εκπαιδεύονται η εκπαίδευση και όλα τα υπόλοιπα μέτρα έχουν πραγματικά αντίκρισμα και αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μειώσουμε το ε, επίπεδο των μικρομεσαίων, των ε, ενδιάμεσων, προκειμένου να διασφαλίσουμε και την ε, χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επίσης από τα αντιευτικά ταμεία, Ζωάννα, διδαχτήκαμε από τα παθήματά μας στο Λίβερπουλ, στο Μάντσεστερ, στο Πρέστον. Υπάρχουν καινοτομικέ εργασίες σε ό,τι αφορά τα κλάστερ για τις καινοτομικέ επιχειρήσεις. Αυτές οι στρατηγικές λοιπόν περιλαμβάνουν τα διδάγματα των ερθωτικών ταμείων. Συμφωνώ απόλυτα με τον Άνταμ σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι κατεπήγον το θέμα αυτό, κατεπήγον το πρόβλημα αυτό και τέλος, αυτό πώς εντάσσεται στη γενικότερη βιομηχανική πολιτική και την πολιτική για την ψηφιακή στρατηγική. Γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει πραγματικά τεράστιο κενό και είναι επονίδιστο αυτό σε ό,τι αφορά τα φύλλα, σε ό,τι αφορά ε, τις εθνότητες, την ε, κοινότητα των μαύρων. Πώς θα διασφαλίσουμε λοιπόν ότι η πολιτική μας θα ενισχύσει την ισότητα για όλους. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενος μιλητής. Ο κύριος Κέλλη. Ίσως ε, να έχει μια διαφορετική διάσταση άποψη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Τζοάννα και την Πατρίσα για τις παρουσιάσεις τους. Νομίζω κάπως αλληλοσυμπληρώθηκαν. Διότι η Πατρίσιο. Είπε ότι οι προθέσει μα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέχουν πολύ από το τι συμβαίνει στην πράξη και κάπω το επενήχθηκε αυτό και η Τζοάννα. Επιχειρηματικότητα λοιπόν. Τι εννοούμε όταν λέμε «μικρομεσές» καταρχά. Είπαμε στην Ιρλανδία κάτω από 50 εργαζομένου. και με όλη την νομοθεσία και τι δοκιμασίε τι οποίε υποβάλλουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα πρέπει να τι διακρίνουμε πρώτα απ' όλα σε διαφορετικέ κατηγορίες. Άλλο οι μεγάλες, άλλο οι μεσαίες, άλλο οι μικρές και άλλο οι πολύ μικρές. Το να μπαίνει το 90% των εταιριών μας στην κατηγορία μικρομεσαίε και να προβλέπουμε τα ίδια για όλους δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Η Τζοάννα ίσω να μπορούσε να σχολιάσει το γεγονός ότι ενώ οι προθέσεις του κόσμου ε, λόγω χάρη και του Horizon ήταν πολύ καλές ε, σκοντάφτει ο, ο το πρόβλημα των ε, διαμεσολαβητών που έλεγε η Πατρίσια τι γίνεται από την κυβέρνηση όμως στην Ιρλανδία τι μπορεί να κάνουν οι κυβερνήσεις για να διευκολύνουν τις μικρομεσαίες και τέλος για το θέμα των δεξιοτήτων είναι κάτι που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μπορεί κάτι να γίνει εδώ, ώστε οι εργαζόμενοι που πάνε στις μικρομεσαίες έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά που υπάρχει, που προσφέρεται. Επίσης, για την νομοθεσία μας είπατε ότι είναι πολλές οι νεοσύστατες στην Ιρλανδία που έχουν περισσότερες πιθανότητες ανάπτυξης φέτος. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριος Μπορέλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύσκολο να επινοήσουμε πολιτικές για τις μικρομεσαίες της Ευρώπης με μια ευρωπαϊκή ενιαία αγορά εφόσον υπάρχει τέτοια διαφορετική φορολογική πίεση μεταξύ των 28 κρατών μελών. Ε, το, το εισόδημα από τους φόρους πολλές φορές Ε, χρησιμοποιείται από ευρωπαϊκές χώρες εφόσον ε, προβλεφθούν ελαφρύνσεις προκειμένου να προσελκυστούν ε, επί που έτσι μετατοπίζονται. Αυτό το έκανε η Ιρλανδία σε μεγάλο βαθμό όπως ξέρουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μήπως πρέπει να αρχίσει σοβαρά να ασχολείται και με το θέμα το φορολογικό των κρατών μελών. Μήπως πρέπει να γίνει και αυτό ένα αναπόσπαστο τμήμα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ευχαριστούμε κυρία Σαντέρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα σχόλιο και μια ερώτηση. Καταρχάς, να χαιρετήσω τις προσπάθειες που έχουν γίνει και τις πολύ καλές προθέσεις, όπως βλέπουμε όλων. Όμως, στην πράξη, επιχειρήσεις, όπως βλέπετε, δεν... Ε, οι καλές προθέσεις δεν αρκούν ε, ιδίως για τις μικρομεσαίες, υπάρχει πραγματικά ένας αγώνας δρόμου. Ε, αγώνας δρόμου για να βρουν πρώτα απ' όλα τις σωστές πληροφορίες, καμιά φορά στον ιστότοπο, σε ιστότοπο του δικτύου, αλλά αν είναι στα αγγλικά μπορεί να μην γνωρίζουν τη γλώσσα. Μετά για να βρουν τον κατάλληλο συνομιλητή, τον κατάλληλο χρηματοπιστωτικό ε, μεσάζοντα, για να βρουν τα κονδύλια που προβλέπονται από τα διάφορα προγράμματα, μετά να ετοιμάσουν τα, τους φακέλους υποψηφιότητας, παν, όχι πάντοτε εύκολο, μετά να περάσουν από ελέγχους που πολλές φορές είναι ιδιαίτερα αυστηροί, δαπανηροί για τις εταιρείες Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που ήθελα να κάνω. Τα πράγματα παραμένουν πάρα πολύ περίπλοκα για τις μικρομεσαίες παρά την καλή βούληση που επαγγελιζόμαστε ότι έχουμε. και τώρα μια ερώτηση προς την κυρία Ντρέκ Είπατε ότι το ποσοστό ανανέωση των επιχειρήσεων φτάνει είναι σταθερό μάλλον, είπατε, στα πλαίσια του Horizon 2020 και ότι πολλές νέες επιχειρήσεις θα ε, εμφανίζονται ήδη σε αυτό το πρόγραμμα. Εγώ θα ήθελα περισσότερα στοιχεία για τις επιχειρήσεις που ήδη έχουν υποστηριχθεί. Έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν αυτή την στήριξη, να ξανακάνουν αίτηση, ή τι έχει αποθαρρύνει μια δύσκολη πρώτη εμπειρία ενδεχομένω οπότε δεν θα το κάνουν καν. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάνκα, ευχαριστούμε. Είδαμε ότι σε καιρό κρίσης τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είδα και εγώ με τα μάτια μου τι έγινε με αυτή τη σαπουνόφουσκα πόλο και μεγάλωνε και διωγγωνόταν και τελικά έσκασε. Ε, αυτοί που επιβίωσαν ήταν, αυτοί που οι πλέον ευέλικτοι. Και είδαμε ότι ο ε, επιχειρηματία που τα κατάφερε ήταν αυτό που είχε θετική στάση στα πράγματα. Πολλέ φορέ η θετική σκέψη κάνει όλη τη διαφορά. Για αυτά που είπε λοιπόν το κύριο Ρούμπικ, είναι σημαντικό στο τέλο μια χρονιά να έχει κάποιο κέρδο μια επιχείρηση ε, Βέβαια, πρέπει να υπάρχει και ρευστότητα, διότι στα χαρτιά μπορεί κανείς να παρουσιάζει κέρδος, αλλά πρέπει να υπάρχει και στην τράπεζα κάτι. Για μας λοιπόν ε, έχουμε εγκρίνει πολλά νομοθετήματα, όμως ε, ένα σημαντικό στοιχείο είναι η εγκύρη πληρωμή των επιχειρήσεων μέσα σε 30 μέρες. Βλέπουμε για τον επιχειρηματικό κόσμο προβλέπονται 62 μέρες το πολύ στην Ιρλανδία. Πώς το, ε, προβλέ... το αντιλαμβάνεστε το θέμα αυτό στη χώρα σας για τις χρηματοδοτήσεις. Πιστεύετε ότι προβλέπονται αρκετά για να προχωρήσουν και να συνεχίσουν να λειτουργούν οι εταιρείε. Ευχαριστούμε η κυρία Κάπελ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις δύο κυρίες για τις παρουσιάσεις τους, ιδιαίτερα στην κυρία Τρέκη, η οποία μίλησε για το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τόνισε την πολύ σημαντική διάστασή τους, γιατί όλοι ξέρουμε τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά το 99% του ιδιωτικού κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο τρίτα των απασχολούμενων στον δυτικό τομέα απασχολούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επίσης μεγάλο τμήμα των φορολογικών εσόδων προέρχεται από μικρομεσαίες επιχειρήσεων. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει η πολιτική έντονα να ασχοληθεί με το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα πρέπει, το δείξατε άλλωστε κυρία Ντρέικ, να απαντήσουμε οι συνθήκες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην έχουν χρέη, να έχουν κέρδη. Μείωση λοιπόν της γραφειοκρατίας, το αναφέρεται ότι θα υπάρχουν και θα πρέπει να υπάρξουν σχετικά μέτρα και υπάρχουν διάφορες συστάσεις σαν χώρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Θα κάνετε όμως προτάσεις για το πώς, θα κάνετε και εσείς προτάσεις για το πώς μειώνεται η γραφειοκρατία σε ό,τι αφορά τα εμπορικά εμπόδια που επίσης θα πρέπει να μειωθούν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ύστερα, κυρία Κάλλον, μιλήσατε για την πρόσβαση στις πιστώσεις. Ε, το πιο σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κόσμε, Ορίζον 2020, πολύ σημαντικά προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας παρακαλώ λοιπόν και σας ρωτώ όπου ο το ανέφερε, τις αφορολογητές ζώνες στην ε, Γαλλία. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει, να αποτελεί μια βέλτιστη πρακτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς αξιολογείται λοιπόν το μέτρο αυτό της Γαλλίας και μια δεύτερη προσθήκη, τα ενισχυμένα κλάστερ Έχουμε κάποιες εμπειρίες. Θα μπορούσε και αυτό να αποτελέσει λοιπόν βέλτιστη πρακτική για την προώθηση μικρών επιχειρήσεων και για την μείωση της γραφειοκρατίας. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Μαρτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω για την έμφαση που δώσατε στι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, γιατί παίζουν πραγματικά ένα ρόλο εξαιρετικά σημαντικό. Μια ερώτηση, γιατί άκουσα κάποια πράγματα που με ενοχλούν κάπω. Διότι εάν θέλουμε ανάπτυξη και μείωση του κόστου εργασία, μείωση των φόρων, μείωση τη νομοθεσία, μείωση του εργασιακού καταστατικού, ε, ε, δεν είναι πολύ καλό αυτό που θα πετύχουμε στην Ευρώπη θα είναι πάρα πολύ καλό για να μπορέσουν να μεγαλώσουν κι άλλο και να αναπτυχθούν οι εξτρεμισμοί, οι ακραίε τάσει. Λοιπόν, για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, σα λέμε τα, τα σίκα σίκα και τι σκάφη σκάφη. Ποιο είναι ο ρόλο των τραπεζών σε αυτή την κρίση. Στη Γαλλία το παιχνίδι του ήταν βρώμικο. Ε, ουδέποτε δεν ε, δέχτηκαν τη χρηματοδότηση των ε, μικρών επιχειρήσεων. Έτσι. Δεν ικανοποίησαν τα αιτήματά του και πολλέ πτώχευσαν για αυτόν τον το λόγο. Και έπειτα για τι πολυεθνικέ, τι πολύ μεγάλε εταιρείε που απασχολούν ε, και συνεργάζονται με, πολύ, με πολλές πολύ μικρές επιχειρήσεις. Πολλές φορές αυτές εξασφαλίζουν τη λειτουργία του μεγάλου ομίλου και πολλές φορές καθυστερούν πληρωμές 80 και 100 μέρες. Γιατί για να πάρει η μικρή εταιρεία τη σύμβαση πρέπει να δεχτεί αυτόν τον όρο. Εκεί λοιπόν πρέπει να ε, καταγγείλουμε την υπεργολαβία διότι είναι υπεύθυνη για πολλές πτωχεύσεις. Και έπειτα για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τη σωστή τους διάκριση. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά για τα κλάστερ, και εδώ θα θέλαμε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι κλάστερ μεταξύ μικρών επιχειρήσεων είναι πολύ καλή ιδέα. Αλλά πρέπει να... Ε, διαδοθούν και οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Πρόσφατα είχα την τύχη να πάω στο βορρά της Ιταλίας επίσκεψη και να δω τι μέσα έχουν για την καλή εμπορία, διαφήμιση, την ε, προώθηση των προϊόντων τους. Είναι πιο, δυνα... Ε, πιο δυνατός κανείς όταν ε, εργάζεται σε ομάδα, ενισχύσει τη ενώση για να προωθήσει τα προϊόντα του, αλλά και για την πρόσβαση στις πληροφορίες των μισθωτών των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Αυτή είναι συνήθως η φτωχή συγγενής της νομοθεσίας ή της πρόσβασης τέλος πάντων στην νομοθετική πληροφορία. Και για αυτούς κάτι να κάνουμε. Ευχαριστούμε. Τελευταίος ο μιλητής, ο κύριος Μαραγκάλ. Και μετά την παρέμβασή του θα ζητήσω από εσάς να απαντήσετε. Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θέλω να σας πω ότι συμβαίνει στην Καταλωνία, στην Ισπανία. Έχουμε επιχειρηματική δομή πολύ συγκεκριμένη και όλα αυτά συμφωνούν με μέρος της ομιλίας σας, αλλά όχι με όλη την ομιλία σας. Έχουμε διαφορετική, υπάρχει διαφορά δυστυχώς αρνητική από πλευράς φορολογικής μεταχείρισης και υπάρχουν και τρία άλλα στοιχεία. Πρώτον, η πρόσβαση στη πίστοση. Δεύτερον, το κόστος της ενέργειας. Και είναι διπλάσιο το κόστος ενέργειας για μας σε σχέση με τις άλλες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άρα υπάρχει πολιτική ευθύνη και κρατική ευθύνη και περιφερειακή ευθύνη. και η Ευρώπη πρέπει να δράσει σε αυτό το τομέα. Ε, βάση μεγέθους δεν θα έπρεπε να μιλούμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά μόνο για μικρές, μόνο small. Και πρέπει να υπάρχουν ενισχύσεις για να αυξήσουν το μέγεθός τους οι επιχειρήσεις αυτές. Οφείλουμε να επενδύσουμε περισσότερα στην επαγγελματική εκπαίδευση και στην κατάρτιση και στο να συνδέσουμε αυτού του είδους τις μορφές εκπαίδευσης με τον παραγωγικό ιστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Ο διάβλος επικοινωνίας δεν έχει ανοίξει, διότι οι επιχειρήσεις οι μικρομεσαίες είναι διάσπαρτες και είναι και μικρές το δέμας και δεν ξέρουν που βρίσκεται το εκάστοτε κέντρο κατάρτισης. Πρέπει λοιπόν να τους φέρουμε πιο κοντά. Από εκεί και πέρα, το σχέδιο το επενδυτικό πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, ο λόγος, οι αναλογίες δεν είναι ικανοποιητικές του πόση προσοχή δίνεται στις μεγάλες υποδομές από τη μία και στις μικρομεσαίες, μικρές δηλαδή επιχειρήσεις από την άλλη. Σε τοπικό επίπεδο πρέπει να είμαστε πιο ενεργητικοί και να έχουμε όλους τους μηχανισμούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και να ζητήσω από την κυρία Τζοάν Αντρέικ, η οποία είναι από τη Μάλτα, σπούδασε στη Μάλτα και ήταν και η επικεφαλής της ε, αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Μάλτα. νομίζω είστε πολύ έμπειροι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα σχετικά θέματα. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις ερωτήσεις, για το ενδιαφέρον σας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να απαντήσω μόνο στις βασικές ερωτήσεις, μόνο στο νόημα αν θέλετε όλων των ερωτήσεων που μου θέσατε. Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να επεκταθώ αρκετά. Ε, επιτρέψτε μου όμως να ξεκινήσω με, το, με την πολύ θεμητή κριτική της Πατρίσια ε, σε σχέση με τα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία, με την διάρθρωσή τους μέσω των διαφόρων τραπεζών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υφιστάμενων και μη, ίσως δεν είναι όργανα αυτά που θα βγουν έξω στην αγορά επιτόπου για να αρχίσουν να αναζητούν ε, επιτακτικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις οποίες να βοηθήσουν. Υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση στις τράπεζες να υποβάλουν αίτηση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για να πιστοποιηθούν αν θέλετε οι ίδιες οι τράπεζες ότι δηλαδή μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά ε, μέσα ε, στη δικιά τους αν θέλετε περιφέρεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμείς ε, δουλεύουμε με τη νέα γενιά του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων το οποίο μετά από 20 χρόνια ε, θα έχει νέους ε, επικεφαλής ε, στις υπηρεσίες του από τον Ιανουάριο του 2015. Είναι μια εταιρική σχέση αυτή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των επιχειρηματικών οργανώσεων, των υπηρεσιών και φορέων που δουλεύουν υπέρ της ανάπτυξης. Συνεργαζόμαστε δηλαδή στενά με όλους όσοι είναι κοντά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να έχουν αυτές περισσότερες δεξιότητες, περισσότερες ικανότητες για να μπορούν να διεκδικήσουν και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Και το, το πιο σημαντικό είναι να μεριμνήσουμε ότι οι τράπεζες θα κάνουν μια σωστή αξιολόγηση κινδύνου των έργων που υποβάλλουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες από μόνες τους δεν μπορούν να αναλάβουν όλο αυτό το ε, ε, βάρος των κονδυλίων. Θα ήθελα λοιπόν να δράξω αυτή την ευκαιρία για να δηλώσω ότι και εμείς πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα, να εκπαιδευτούμε καλύτερα, να μάθουμε περισσότερα για τις τράπεζες και να είμαστε σίγουροι ότι οι τράπεζες έχουν εκπαιδευτεί καλύτερα για να κάνουν καλύτερη και πιο δίκαιη αξιολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ως προς το νομοθετικό άχθος και υπήρχε τις ερωτήσεις για την περιβαλλοντική νομοθεσία. Κοιτάξτε, το να απαλλάσσονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την υποχρέωση τήρησης ορισμένων νομοθετικών διατάξεων δεν είναι κάτι που ε, επιθυμούν ούτε καν οι ίδιες. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κάνουμε το παν με τη βοήθεια του Γενικού Γραμματέα έτσι ώστε να βοηθήσουμε και τις άλλες υπηρεσίες μας που δεν εστιάζουν τόσο πολύ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο εμείς, να τα έχουν υπόψη τους όλα αυτά. Δηλαδή, όταν φτιάχνουν οι άλλε υπηρεσίε νομοθεσία, π.χ. περιβαλλοντική, να έχουν υπόψη του τον αντίκτυπο που αυτή θα έχει στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Η αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών τη αξιολόγηση αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι 27 Νοεμβρίου παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και, το οποίο και υιοθέτησε και ψήφισμα σχετικό ε, για ε, την αξιολόγηση αντικτύπου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά είναι σημαντικά, διότι γίνεται ακόμα πιο σοβαρή η αξιολόγηση αντικτύπου και ακόμα πιο ε, στέρεα σαν κείμενο δεν μπορεί πλέον να παρακαμφθεί. Έχουμε Σοβαρέ κατευθυντηρίες γραμμέ, οι οποίε εφαρμόζονται σωστά και αυτό πρέπει να γίνεται. Από εκεί και πέρα, μέσω του προγράμματο REFIT για την αναδιαμόρφωση τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. όποια νομοθετική διάταξη είναι απειρχαιωμένη, δεν ταιριάζει καλά, θα πρέπει να διαγραφεί, θα πρέπει να φύγει. χάρη σε αυτό το πρόγραμμα θα τα καταφέρουμε αυτά με το πρόγραμμα REFIT. Ε, της αναμόρφωσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε και όχι να απαλλάσσουμε τη χύψη μικρομεσαία επιχείρηση από την υποχρέωσή της να συμμορφώνεται με τον νόμο και να τον τηρεί. Θέλω να σας μιλήσω και για το ε, πράσινο σχέδιο δράσης. Στόχος είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να έχουν τη δική τους ευκαιρία με ίδιους πόρους, δηλαδή να βρουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στις πράσινες αγορές. Και άρα εμείς δουλεύουμε με τους εμπλεκόμενους φορείς στην πράσινη οικονομία, με τις πράσινες αγορές, έτσι ώστε να δρομολογούνται οι δράσεις, να γίνεται αξιολόγηση του αντικτύπου. Για παράδειγμα, παρατηρητήριο αποδοτικότητας πόρων έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μάθουν πόσο αποδοτικές είναι από πλευρά των δικών τους πόρων και πώς μπορούν να τα βελτιώσουν αυτά και πώς μπορούν να μπουν στην πράσινη αγορά. Ως προς το ε, κεφάλαιο κινδύνου, να αναφερθώ στο πρόγραμμα COSME. Ναι, λείπουν τα κεφάλαια αυτά. Να θέλει δηλαδή κάποιος να βάλει χρήματα αναλαμβάνοντα το ρίσκο. Προτείνουμε στο Small Business Act διαβούλευση να χτιστεί και να αναδομηθεί η αγορά των venture capital, των επενδυτικών κεφαλαίων μέσω σύμπραξης. Όλα αυτά, το κόσμο, δίνουν μια βιώσιμη ευκαιρία. Τα χρήματα μπορεί να είναι λίγα, όμως αυτά λειτουργούν ως μόχλευση. 21 ε, δις ευρώ τελικά μοχλεύθηκαν. Ε, για ένα ευρώ που μπήκε ε, στο πρόγραμμα ως επένδυση, άλλα 30 ευρώ μοχλεύθηκαν και κινητοποιήθηκαν και βρέθηκαν τελικά. αυτό είναι πολύ θετικό. Προσαρμόσαμε τους κανόνες του κόσμου για να έχουμε περισσότερους ιδιώτες επενθυτές και έχουμε και την επερχόμενη Ένωση των Κεφαλαιακών Αργορών. Και αυτό θα είναι πολύ θετικό για το πρόγραμμα COSME. Σίγουρα πρέπει να ε, εστιάσουμε την προσοχή μας όλα αυτά και με βάση το νέο SBA, το Small Business Act. Ε, χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για όλα αυτά. Είχαμε πολύ καλό feedback, ανατροφοδότηση για το ποιο αντίκτυπο είχαν οι πράξεις μας αλλά χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο. Το 70 80% των πραγμάτων που κάνουμε την χάνει ευρεία συστήριξης. Τώρα, ε, από, την, ε, από τους χρήστες και τους αποδέκτες. Τι κάνουμε για τις χώρες του Νότου. Κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Απαντώ. Έχουμε την πρωτοβουλία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. SME Initiative δοκιμάζεται ακόμα, την εξετάζουμε. Είναι πρόσκληση προς τα κράτη-μέλη κάποια από τα διαρθρωτικά του ταμεία να τα αφιερώσουν σε αυτή την κατεύθυνση μαζί με τα χρήματα που έρχονται από τα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία, έτσι ώστε να υπάρξει επένδυση σε στρατηγικές επενδύσεις και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το σχέδιο ε, Juncker με το νέο Ταμείο Επενδύσεων πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση επίσης. Και ε, πληροφοριακά λέω ότι η συμμετοχή στα χρηματοδοτικά εργαλεία ΣΥΠ από τις χώρες του Νότου π.χ. έρχεται σε μεγαλύτερο βαθμό από την Ιταλία και την Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν και όλα αυτά θα παρθούν, θα ληφθούν, αν θέλετε, από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τι σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2016. Να απελευθερώσουμε το δυναμικό στις αναδυόμενες βιομηχανίες, να τροποποιήσουμε την αλυσίδα μέσω της οποίας δημιουργείται προστιθέμενη αξία να ενισχύσουμε τη διασυνοριακή περιφερειακή συνεργασία με τα κλάστερ. Με τις συστάδες αυτές τις επιχειρηματικές πάντοτε το αποτέλεσμα είναι η κοινοτομία. Οι μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις λειτουργούν μαζί δίπλα-δίπλα και ε, τροφοδοτεί η μία την άλλη. Οι δεξιότητες, τα προσόντα, οι ικανότητες είναι προτεραιότητα στο νέο SBA, Small Business Act και ε, το επικοινωνιακό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Δεν περηφανευόμαστε ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε 23 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται και λειτουργούν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Όμως, προσπαθούμε να διαδώσουμε όσο δυνατόν περισσότερο την πολιτική μας και έχουμε και τις συμβουλευτικές ε, υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού Δικτύου. Και πρέπει να λειτουργήσουν ως προωθητήρες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επί τόπου με τη δική μας στήριξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Κάλαν. Η Πατρίσια ήταν ε, η επιχειρηματίας του 2007 έλαβε το σχετικό βραβείο και έχει λάβει και άλλα βραβεία, συμμετέχει σε πανεπιστήμια, ιδρύματα και στην Ιρλανδία έχει βραβευθεί και στην ε, ε, Επιτροπή Επιχειρηματιών του Business Europe. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα και εγώ να ομοτοποιήσω τις απαντήσεις. Να ξεκινήσω από την παραγωγή και το, την έννοια των κλάστερ, γιατί όπως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είχαμε κινηθεί πιο πολύ ε, στις υπηρεσίες και τώρα εστιαζόμαστε πιο πολύ στην παραγωγή. Νομίζω ότι είναι κρίσιμη σημασία να κινούνται όλα από τις επιχειρήσεις. Στην Ιρλανδία υπάρχει μια οργάνωση που εκπροσωπεί όλες τις επιχειρήσεις και εμείς είμαστε ηγετικό, ηγετικοί. Είμαστε λοιπόν άτομα που παράγουν και θέλουμε να ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές και όλα αυτά θέλουμε να περνούν και στις κυβερνητικές στρατηγικές. Άρα υπάρχει ευθύνη και στις επιχειρήσεις να ηγηθούν του τι γίνεται. Η χώρα μας ευτυχώς είναι μικρή. Και πάλι λοιπόν οι πολυεθνικοί όμιλοι φαίνεται ότι εστιάζονται σε κάποιες συγκεκριμένες πόλες ε, ε, ICT, οι επιχειρήσεις αυτές είναι σε συστάτες, σε κλάστερ και είμαστε λοιπόν είμαστε πολύ ενεργοί και ενθαρρύνουμε λοιπόν το προσωπικό να δραστηριοποιηθεί. Χρειάστηκε λοιπόν να υπερπηδήσουμε διάφορα θέματα για την πνευματική ιδιοκτησία, αλλά αυτό έγινε με πολύ δημιουργικό τρόπο. Είναι καλό λοιπόν οι εργάτες, οι εργαζόμενοι στις πολυεθνικές να κάνουν σχόλια και αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο με μεγάλη μας χαρά θα το μοιραστούμε με άλλους. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και τις επιδοτήσεις τώρα, οι επιχειρήσεις δεν πιστεύουν ότι αυτό έρχεται από το κόσμο ή από άλλα προγράμματα σε επιχειρησιακό επίπεδο. Θεωρούν ότι αυτό προέρχεται από κυβερνητικό επίπεδο και ότι υπάρχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την παραγωγή από ότι για τις υπηρεσίες. Γιατί είναι πιο ακριβή και η σύσταση υποδομών για την παραγωγή σε ό,τι αφορά τώρα θέματα νομοθεσίας. Και πάλι έγινε ένα εργαστήριο αυτή την εβδομάδα, ήρθαν εκπρόσωποι του ΆΣΑ των συναδέλφων από τον Εμένο Βασίλειο. Είμαστε λοιπόν πολύ ευγνώμονες για αυτό που συνέβη στην ΕΜΒΗ. Υπάρχουν πραγματικοί στόχοι, πραγματικές κυρώσεις, πραγματική εφαρμογή της καλής νομοθεσίας και οι κυβερνήσεις αυτό το διαδίδουν. δεν κοιτάμε καν θέματα νομοθεσίας μακροοικονομικής. Αποδεχόμαστε το γεγονός ότι υπάρχει νομοθεσία. Προσπαθούμε λοιπόν να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν την νομοθεσία. Καταλαβαίνετε, αν είναι πιο απλό να συμπληρώσει κανείς ένα έντυπο, το κάνει πιο εύκολα. Και εκεί νομίζω ότι οι επιχειρήσεις ε, νιώθουν τον αντίκτυπο. Όχι, δεν πρόκειται να καταργήσουμε το εργασιακό δίκαιο, αλλά έχουμε για παράδειγμα μια νομοθεσία για το ωράριο, για τις ώρες εργασίας. Μία επιχείρηση λοιπόν πρέπει να συμπληρώνει μία φόρμα κάθε εβδομάδα για κάθε υπάλληλο. Ακόμα και τα γραφεία που χρειάζονται για την αρχιοθέτηση είναι προβληματικά για τόσο, πολύ, τόσο πολλά έντυπα. Υπάρχουν λοιπόν εύκολοι τρόποι να διευκολύνουμε τη ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις καθυστερημένες πληρωμές. είναι το ερώτημα που τέθηκε αυτό. 62 ημέρες ε, είναι η προθεσμία στην Ιρλανδία, αλλά ασκούμε πίεση στην κυβέρνηση να βοηθάει τις επιχειρήσεις, δίνοντας το καλό παράδειγμα. Άρα, σε 15 ημέρες λοιπόν ζητούμε να πληρώνονται τα χρέη και οι τράπεζες. Μπορεί να γίνει λοιπόν αυτό, ακόμα και αν υπάρχουν άλλε προτεραιότητε. Αν υπάρχει δέσμευση στην παρούσα φάση, γίνεται μια συζήτηση για το κατά πόσο θα πρέπει το, η προθεσμία αυτή να είναι 30 ημέρε, αλλά πολλέ επιχειρήσει ε, έχουν συμβάσει που προβλέπουν μεγαλύτερε προθεσμίε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υποχρεωτικά θέλουμε 30 ημέρε προθεσμία στην Ιρλανδία. Είναι πολύ μικρό, μικρή οικονομία. Αλλά αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίσει την προθεσμία των 30 ημερών. Θα το αποδεχόταν ε, όλος ο κόσμος, οι πολυεθνικές. Θέτετε ερωτήματα, γιατί δεν μπορεί κανείς να λαμβάνει αποφάσεις, επαναλαμβάνω, σε επίπεδο χώρας. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας. Αλλά αυτό θα χρειάζεται για να λύσουμε τα προβλήματα. Βέλτιστες πρακτικέ, κώδικας, συντελογίας, αλλαγή της κουλτούρας. Αλλά το θέμα είναι το τι θέλουμε να εφαρμόσουμε, τι σκοπό έχουν τα μέτρα σε ό,τι αφορά τα προσόντα, τη βάση των ικανοτήτων. Θεωρώ ότι αυτό πραγματικά θα πρέπει να το ορίσει η οικονομία. Η κυβέρνηση δεν ξέρει τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση και τον μηχανισμό χρηματοδότησης που υπάρχει. Οι ομάδες και τα κλάστερ των επιχειρήσεων ε, συνέρχονται, δημιουργούν αυτό το skill net, το δίκτυο ικανοτήτων, το οποίο και χρησιμοποιείται για να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους και τους ανέργους. Αλλά μιλάμε για μικρή χρηματοδότηση, μικρό κεφάλαιο, μικρό κονδύλι σε σχέση με τις άλλες ε, οργανώσεις που εκπαιδεύουν τα άτομα χωρίς να ξέρουν όμως τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Πολύ απλά δεν γνωρίζουν τα δεδομένα που είναι άγνωστα σε αυτούς και αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο μήνυμα σε ό,τι αφορά την αποτυχία. Πρόσφατα αλλάξαμε την ομοθεσία μας για τα τρία έτη πτώχευσης από 12 χρόνια. Ήταν σημαντικό αυτό, αλλά εδώ χρειαζόμαστε πολύ πιο ενεργά μέτρα για προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας. να αναπτύξουμε την οτροπία ότι η αποτυχία είναι κάτι από το οποίο θα πρέπει να διδαχθούμε. Στην Ιρλανδία, ειλικρινά, ο κόσμο είναι ενθουσιασμένο όταν κάποιο αποτυχάνει. Θα πρέπει να υπάρχουν νομοθετικέ διαδικασίε και θα το, θυμάται ο κόσμο αυτό για πολλά χρόνια. Υπάρχει λοιπόν πολλή δουλειά να γίνει σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό και αν θέλει πραγματικά κανείς να είναι ανταγωνιστικός, πολύ απλά υπάρχει και το ενδεχόμενο της αποτυχίας. Είναι τμήμα του συστήματος. Του θεωρώ ότι δεν έχει λάβει τη σωστή προσοχή όμως το θέμα αυτό. Για την επιχειρηματικότητα μεταξύ των μειονοτήτων. Και πάλι είδαμε ότι τα στοχευμένα προγράμματα για τις γυναίκες, για συγκεκριμένες αθνοτικές μειονότητες, Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι τα άτομα αυτά που είχαν ε, συμμετάσχει στα προγράμματα, στα αρχικά, σε αρχικές φάσεις ήθελαν κάτι συγκεκριμένο. Συχνά αυτό αποτελεί, ξέρετε, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό με το οποίο ταυτίζεται κανεί ότι είναι γυναίκα, ότι ανήκει σε μια εθνική μειονότητα. Αλλά στην τελική ανάλυση ο κόσμο αυτό θέλει να ενταχθεί στο mainstream. Θέλει να γίνει όπω όλοι οι υπόλοιποι και να βρουν δουλειέ. Και υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα προγράμματα χρηματοδότηση για τι ε, ειδικέ αυτέ ομάδε. Και σε αυτέ συγκαταλέγονται και οι νέοι. Οι βέλτιστε πρακτικέ. Κάθε καλή πολιτική που προτείνουμε και προσπιζόμαστε. υπάρχει και κάπου αλλού στην Ευρώπη. Αλλά η επικοινωνία είναι πάρα πολύ δύσκολη σε ό,τι αφορά τι μικρέ επιχειρήσει. Δεν σα ζηλεύω καθόλου. Αλλά πιστεύω ότι χρειάζεστε τις σωστές πληροφορίες. Ιστοσελίδες. Μπήκα λοιπόν στην ιστοσελίδα του κόσμου. Προσπάθησα να βρω πληροφορίε για τη χώρα μα. Και πολύ απλά δεν τι βρήκα τι πληροφορίε αυτέ. Άρα χρειαζόμαστε τα βασικά στοιχεία να λειτουργούν καλά. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την φορολογική πολιτική, κάθε χώρα και κάθε κυβέρνηση, πολλά ακούμε για το τι συμβαίνει στην Ιρλανδία, αλλά υπάρχουν και πολλέ πολλές άλλες χώρες που προσφέρουν χαμηλό φορολογικό καθεστώς στις ε, πολυεθνικές και ακόμα σε ό,τι αφορά την ε, έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία, όλα αυτά. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από πλευράς μικρών επιχειρήσεων έχουμε την αίσθηση ότι δεν έχουμε την υποστηρίξη της ε, κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της επιχειρηματικότητας, σε ό,τι αφορά το 3% για παράδειγμα για το κεφαλαϊκό κέρδος, ανεξάρτητα από το αν ένας επιχειρηματίας πουλάει μια επιχείρηση για να ξαναχτίσει μια άλλη επιχείρηση ή όχι. Χρειαζόμαστε λοιπόν ανταγωνιστικότητα και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά τι προλογικέ πολιτικέ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ λέει ο ευχαριστούμε και τις δύο ομιλήτριες για όλες τους τις ε, παρατηρήσεις, για τις ομιλίες σας. Ήταν πραγματικά ιδιαίτερα πλούσιες και επικοδομητικές. Επόμενο τμήμα της ακροασής μας, πρόσβαση των μικρομεσαίων στις πιστώσεις. Ε, δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση. Θα ζητήσω από τον κύριο Γκί Γκέλντοφ να λάβει το λόγο. Μετά την ε, οπτική γωνία των ίδιων των μικρομεσαίων, από δύο διαφορετικές πλευρές ε, της Υπήρου μας, από το βορρά και το νότο, τώρα ε, περνάμε στο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Βέλγιο. Ο κύριος Γκί Γκέλτχοφ αποφύτησε το 1991 από το Business School του Σολβέ, το ελεύθερο πανεπιστήμιο των Βρυξελών. Και είχε έντονη δράση ως επικεφαλής ομάδας επιχειρηματικούς συμβούλους, στην McKinsey και στην Solvay Business Consulting. Είναι γενικός γραμματέας του φορέα για τα κεφάλαια κινδύνου και τις ε, ιδιωτικές επενδύσεις στο Βέλγιο από το 2004 και είναι ιδιαίτερα δραστήριος σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα λοιπόν να λάβετε το λόγο κύριε Γκέλντοφ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να, από τη ναι, αν θέλετε. Ναι, πολύ καλύτερα τώρα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατάρχα. Θα ήθελα να δώσω μια πλατφόρμα ε, σε όσους χρησιμοποιούν κεφάλαιο κινδύνου να μιλήσουν γιατί θεωρώ ότι το κεφάλαιο κινδύνου είναι ένας μακροπρόθεσμος εταίρος νέων, αλλά όχι μόνο νέων επιχειρήσεων, αλλά και παλαιότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως αναπτύσσονται. Είναι σημαντικό να αναπτύσσονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει να, να συστήνονται, αλλά θα πρέπει να αναπτύσσονται κιόλας. Γι' αυτό και χαίρομαι που όλο και πιο πολλές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Κοινοβουλίου για το κεφάλαιο κινδύνου αρχίζουν να ε, γίνονται αντιληπτές, να αναγνωρίζονται από τους ηθήνοντες, τους πολιτικούς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το κεφάλαιο κινδύνου από μόνο του δεν συγκρίνεται με τις τράπεζες ή με άλλα πιστοτικά ιδρύματα το κεφάλαιο κινδύνου, αποτελεί μια ξεχωριστή ομάδα βασικός στόχος τους είναι να παρέχει ε, ισότητα στις επιχειρήσεις. Δεν ε, πρέπει λοιπόν το κεφάλαιο κινδύνου να αντιμετωπίζεται ως τράπεζα. Κάτι άλλο, οι επιχειρήσεις ε, κεφαλαίου κινδύνου επενδύουν στην πραγματική οικονομία. Δεν ε, επενδύουμε σε χρηματοπιστωτικά ε, μέσα, σε περίπλοκα μέσα, περίπλοκα προϊόντα που δημιουργούν προβλήματα και κανείς δεν τα καταλαβαίνει. Όχι, σε πραγματικές επιχειρήσεις, σε πραγματική τεχνολογία, σε πραγματικό κόσμο επενδύουμε. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό το μήνυμα που θα πρέπει να το διαβιβάσουμε. Είναι σημαντικό τμήμα των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων που θα μπορέσουν να είναι οι προαθλητές του αύριο ενδεχομένω. Οι πιστώσει ασφαλώς ε, ε, δίνουν μόχλευση σε χρηματοδότηση δανεισμού αλλά και σε ήπια προγράμματα ε, χρηματοδότησης γιατί πρέπει να υπάρχει ε, επιχειρηματικό κεφάλαιο προκειμένου να μπορέσει κανείς να α, επιβιώσει. Και τέλος, να πω ότι είμαστε μακροπρόθεσμοι επενδυτές. Επενδύουμε σε επιχειρήσεις. Πολύ συχνά από επιχειρήσεις που προήλθαν από μια πανεπιστημιακή επιχείρηση που έχει καλύψει ένα συγκεκριμένο μόνο για παράδειγμα. για εξαετή περίοδο, οχταετή περίοδο. Δεν είμαστε λοιπόν, ε, τα χτυπάμε και φεύγουμε, είμαστε μακροπρόθεσμοι επενδυτέ. Κάποια αριθμητικά στοιχεία δεν θέλω να σας παραφορτώσω γιατί νομίζω ότι έχετε πρόσβαση σε πολλά δεδομένα. Ε, βλέπετε στις αθώνε ε, σας ότι σήμερα οι επιχείρησεις αυτές ο κλάδος μας ε, επενδύει σε περισσότερες από 20.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Κάθε χρόνο επενδύουμε σε 4.000 επιχειρήσεις. Για νέου συσταθήσεις, επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που δεν έχουν συσταθεί ακόμα και επιχειρήσεις που έχουν ήδη συσταθεί και αναπτύσσονται. Και έχω περιλάβει και τις επιχειρήσεις ανάπτυξης. Οι ετήσιες επενδύσεις, μέσος όρος, κατά μέσο όρο, για τα 7 χρόνια έχω υπολογίσει αυτά τα ποσά μετά την κρίση και θεωρώ ότι το επιχειρηματικό κεφάλαιο ή το κεφάλαιο κινδύνου ε, δεν έχει πέσει ιδιαίτερα. Αυτό που έχει μειωθεί σημαντικά, και αυτό δεν είναι καλό, είναι τα ποσά μόχλευσης από 9 δισεκατομμύρια σε 7 δισεκατομμύρια το 2013. Δεν είναι όλες οι εταιρείε κατάλληλες για κεφάλαιο κινδύνου. Έχουμε συγκεκριμένη στόχευση σε ό,τι αφορά την αγορά. Βλέπετε στα μέσα της διαφάνειας ότι πιο πολλές από τις επενδύσεις, τα πιο πολλά χρήματα που επενδύονται στον κλάδο μας είναι ICT, επιστήμες ζωής και τα τελευταία 5-10 χρόνια όλο και πιο σημαντικός είναι ο κλάδος της πράσινης ενέργειας, clean tech, καθαρής τεχνολογίας. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, είναι δύσκολο να βρούμε τα σωστά στατιστικά στοιχεία γιατί υπάρχει αιματοποίηση ανά κλάδο μια επιχείρηση που ειδικεύεται στις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν συμπεριλαμβάνεται απαραίτητα στους υπολογισμού, αλλά είναι σημαντικό και βλέπουμε ότι 90% των επιχειρήσεων μας που υποστηρίζουμε έχουν τέτοια ανάπτυξη. Επενδύουμε επίσης ε, και σε πιο μεγάλες επιχειρήσεις για να τις βοηθήσουμε να περάσουν στο επόμενο επίπεδο. Και τέλος, το κεφάλαιο κινδύνου δεν είναι μόνο μια αρχική επένδυση. Αν επενδύσουμε ένα δισεκατομμύριο σε μια επιχείρηση σήμερα, βάζουμε θέμα δύο δισεκατομμύρια σε επενδύσεις συνεχιζόμενες προκειμένου να υποστηριχθεί η επιχείρηση σε όλον τον κύκλο ζωή τη, γιατί δεν έχει νόημα να δημιουργηθεί μια νέα επιχείρηση, μια μικρή επιχείρηση, αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση και στη συνέχεια τη ανάπτυξή τη. Και αυτό είναι το τμήμα του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε. Δύο σημεία ήδη έχω αναφέρει ότι τα χρήματα του κεφαλαίου κινδύνου δεν είναι ε, χρέος, αλλά αποτελεί μια μόχλευση σημαντική για τις επιχειρήσεις. αυτό που λέμε είναι ότι ε, βοηθάει την προσέλκυση ήπιου χρήματος, ε, πρόσβαση προγραμμάτων κρατικών, ευρωπαϊκών, επιδοτήσεις, επιδοτήσεις, πολύ σημαντικό σκέλος αυτό σε ό,τι αφορά τα θέματα καινοτομία, αυξάνει τη δυνατότητα δανεισμού και πιο σημαντικό προσελκύει επίση τους επενδυτές ε, από το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσελκύουμε λοιπόν επενδυτέ επειδή είμαστε Ευρωπαίοι, προσελκύουμε επενδυτέ από την Ιαπωνία, από τη ΣΥΠΑ. Χρειάζεται λοιπόν ε, οι τοπικοί ηγετικοί επενδυτέ. Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προσελκύσουμε και τους αλλοδαπούς επένδυτες. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια πραγματικά ζωηρή οικονομία Δεν είμαστε τράπεζε. Όταν πάει κανεί στην τράπεζα και ζητάει λεφτά, τι θα κάνει η τράπεζα. Η τράπεζα θα κάτσει να κοιτάξει κατά πόσον η επιχείρηση αυτή μπορεί να ξεπληρώσει το χρέο τη. Μπορεί να εξυπηρετήσει το χρέο. γιατί φυσικά η τράπεζα δεν θέλει να χάσει χρήματα, να έχει ελληματικούς ισολογισμούς και να δημιουργηθεί ένα παύλος κύκλο από το γεγονός αυτό. Τα κεφάλαια κινδύνου κοιτάνε τους ε, ε, μετόχους και συντονιζόμαστε με τα συμφέροντα της επιχείρησης. Ξέρουν λοιπόν στις πιο πολλές περιπτώσεις τα κεφάλαια κινδύνου την επιχείρηση. Εγώ λοιπόν είμαι στον δικό μου κλάδο εδώ και 20 χρόνια. Ξέρω καλά τον κλάδο και πώς λειτουργεί. Έχουμε μεγάλα δίκτυα επενδυτών, συν επενδυτών που μας συνοδεύουν στις επενδύσεις μας. Και τέλος, χάρη στη γνώση αυτή και την εμπεροπνομοσύνη αυτή, ξέρω ότι αυτό δεν αρέσει πάντα στις επιχειρήσεις που ανοίγουν το κεφάλαιό τους, αλλά δίνουμε συμβουλές, μπορούμε να είμαστε οι κακοί πεθερά αν θέλετε των ε, επιχειρήσεων αυτών, αλλά οι, ακόμα και οι κακές επιθερές πάντα δίνουν ε, συμβουλές προς το συμφέρον των επιχειρήσεων. προκειμένου να τις ε, σπρώξουμε προς την λειτουργική αριστεία. And therefore... Και ως εκ τούτου, Πρόεδρε, αγαπητό κοινό, to see... είναι δραματικό το πώς έχει διαβρωθεί η βάση χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνδυνου τα τελευταία χρόνια. Έχουμε όλο και πιο λίγα χρήματα. Εν μέρει φτάμε κι εμείς. Ως επενδυτές δεν είχαμε την σωστή απόδοση πάντα και κατά μέσο όρο η απόδοση δεν ήταν πάντα τόσο καλή. Αλλά και οι ρυθμιστές και οι πολιτικοί ηθήνοντες δεν μας βοήθησαν. Φυσικά υπάρχει και η ατζέντα η σα και φυσικά θέλετε προστασία των επενδυτών, θέλετε να υπάρχει σταθερότητα στο οικονομικό σύστημα. Όλα αυτά είναι καλά και λογικά. Αλλά ποιες είναι οι συνέπειες, οι μη θελημένες συνέπειες του Solvency 2, του MIFID, όλης της νομοθεσίας. Ποιος τελικά αναλαμβάνει κινδύνους στην κοινωνία. Μία κοινωνία χωρίς κινδύνους. Πολύ απλά αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος ο οποίος θα αναλαμβάνει τον κίνδυνο του επιχειρηματικού κεφαλαίου. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό. Φυσικά υπάρχει χρηματοδότηση από άλλες πήγες. Το δημόσιο χρήμα κινεί την αγορά μέχρι σε ένα βαθμό. Στην Ευρώπη, στην Γαλλία υπάρχουν ε, οργανισμοί. Αν αποφασίσουν να δώσουν χρήματα σε κάποιο ταμείο, μπορούν να κλείσουν τα ταμεία να αποφασίσουν ποια, ποια ταμεία, ποιες ε, κεφάλαια θα διατηρηθούν και ποια δεν θα διατηρηθούν. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας δώσω κάποιες ιδέε. Εγώ δεν είμαι πολιτικός ευθύνων και δεν υποκρίνομαι ότι είμαι τέτοιο. Αλλά να σας δώσω κάποιες σκέψεις, να τις έχετε υπόψη για το τι πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να διευκολύνουμε, θεωρώ, όλο και πιο πολύ την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη κινδύνων. Τα συμφέροντα των νέων θα πρέπει να υποστηριχθούν σε όλους τους σημαντικούς κλάδους σε κάποιες χώρες έχω όλο και πιο πολύ την αίσθηση ότι οι επιχειρηματίες θεωρούνται ε, απαταιώνες που θέλουν μόνο να κλέψουν κέρδη. Δεν είναι σωστό το πνεύμα αυτό. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά θα πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή την ετροπία. Επιχειρηματικό κεφάλαιο, όπως σας είπα, δεν είμαστε τράπεζες και θεωρώ ότι πρέπει να μας μεταχειριστείτε με διαφορετικό τρόπο. Και τέλος, τελευταίο σημείο μην μας σπρώχονται μόνο στα χέρια των δημοσίων επενδυτών. Οι θεσμικοί επενδυτές, οι τράπεζες, οι ασφαλίσεις μπορούν να δίνουν ακόμα και ένα μικρό ποσοστό και να δώσουν τεράστια όθηση στον κλάδο και έχει το πλανέκτημα αυτό ότι πρόκειται για ιδιωτικό χρήμα, το οποίο είναι πολύ πιο θετικό από το να αποφασιστεί κάτι σε ό,τι αφορά τις δημόσιες δαπάνες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για αυτή την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ο Όλιβερ Γκάιντα είναι και αυτός από το Βέλγιο, είναι συνειδητή και πρόεδρος του δικτύου για το crowdfunding στο Βέλγιο και έχει εργαστεί για το κεφάλαιο κινδύνου, τα, την, τις μικροπιστώσεις και την κοινωνική επιχειρηματικότητα και σε ε, εμπορικά και σε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είστε πρώην δημοσιογράφος επίσης ε, από την πλευρά λοιπόν της ε, προβολής και της πληροφόρησης άριστα. Έχετε αποφοιτήσει κι εσείς από το Solve Business School και έχετε σπουδάσει και στη Γερμανία και στο Λονδίνο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε και που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσω. Τα περισσότερα έχουν ήδη υποθεί, αλλά θα προσθέσω μερικές λεπτομέρειες. Ο πρόεδρος Μπούζεκ ανέφερε το πρωί ότι συζητούμε λίγο την αποτυχία των πολιτικών ηθινόντων που 20 χρόνια προσπαθούν και δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Ε, βλέπω ότι και άλλοι είναι εδώ, όπως ο καθηγητής Ρούμπικ που ήταν ε, παρόν και στην αναθεώρηση της στατικής της Λισαβόνας και είδαμε τι επιτυχία επιδιώχθηκε και τι ε, καταφέραμε να έχουμε σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως λοιπόν είναι τώρα μια ευκαιρία εν ώψη της ενδιάμεσης αναθεωρήσης στρατηγικής του 2020 να αναλάβουμε κάποιες δράσεις. Είναι πάντως ε, τουλάχιστον ενθαρρυντικό ότι ένα τρίτο των μέλων αυτής της Επιτροπής είναι εδώ σήμερα για να ακούσουν τι έχουν να πούν 50% ε, των παραγωγών του 60-70% όλων των θέσεων απασχόληση της Ευρώπης και 90% όλων του ΑΕΠ της Ευρώπης. Να πώς θα προωθήσετε τις προτεραιότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, να πώς θα δοθεί όθεση σε όλα αυτά. Πρόσβαση στις πιστώσεις των μικρομεσαίων λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για το crowdfunding. Αν και ο κύριος Γκέλτγοφ ήδη σχολίασε κάποια ζητήματα. Έχουμε εδώ δύο επίπεδο, τη ε, αγορές κεφαλαίων για το επιχειρηματικό κεφάλαιο, για, το, για τα δάνεια, για τις τράπεζες, εάν δουλεύει κανείς σε μια επιχείρηση, ξέρει ότι ε, υπάρχει το ισοζύγιο, το ε, και στα ενεργητικό στα στοιχεία του ενεργητικού βάζουμε το δάνεια, ενώ στα ε, στοιχεία του αποθετικού το επιχειρηματικό κεφάλαιο. Ξέρετε όμως ότι όσα προβλέπονται στην ρευστότητα δεν διατίθενται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκτός να φτάσουν τα 50 εκατομμύρια συναλλαγές και είναι πολύ δύσκολο οι, κεφαλές, οι αγορές κεφαλαίων να χρηματοδοτήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επόμενη δυνατότητα είναι το κεφάλαιο κινδύνου. Αλλά είδαμε πόσο δύσκολος είναι αυτός ο κλάδος. Και μετά η επόμενη λύση είναι οι επιχειρηματίες που στηρίζουν άλλες επιχειρήσεις, οι οποίοι όμως πέφτουν στις άλλες δύο κατηγορίες, έχουν πολύ αυστηρούς κανόνες, δεν μπορούν ελεύθερα να επενδύσουν στις μικρομεσαίες. Εάν συνδυάσουμε αυτούς τους, ε, αυτές τις δύο ομάδες με τις 10 εκατομμύρια μικρομεσαίες που έχουν λιγότερους από 200 εργαζομένους και χρειάζονται κεφάλαια, φτάνουμε τις 10.000 εταιρείες ετησίως το πολύ τα στατιστικά στοιχεία μπορεί να μην είναι σωστά, αλλά επενδύονται 10 δις ευρώ στις μικρομεσαίες ετησίως. Δεν μπορείτε να μου πείτε ότι έχουμε 20 εκατομμύρια μικρομεσαίες στην Ευρώπη που μπορούν από αυτές τις επενδύσεις να επιβιώσουν. Εάν το πιστεύετε, θα έλεγα ότι είστε ανόητοι. Ε, πρέπει να υπάρχει και άλλη πηγή κεφαλαίου. Κάποιος πρέπει να χρηματοδοτήσει τις εταιρείες μας τα κεφάλαια κινδύνου δεν σας δίνουν λεφτά εάν θέλετε να, αν πείτε ότι θέλετε να ιδρύσετε μια εταιρεία. Μόλις έχετε ήδη ένα business plan και κάποιο προϊόν, τότε θα σας χρηματοδοτήσουν. Όλοι αυτοί θα χρηματοδοτήσουν 20 εκατομμύρια μικρομεσαίες, αυτοί που ονομάζουμε φίλοι, οικογένεια και συγγενείς που βάζουν υποθήκη το σπίτι τους, που παίρνουν τα ωφέλη από την κοινωνική τους ασφάλιση και διακινδυνεύουν όλη τους τη ζωή, α, ε, τις οικογένειές τους ακόμη, για να ε, κυνηγήσουν το όνειρό τους. Αυτοί μπορεί να δώσουν μια λύση, αλλά συνήθω αποτυγχάνουν οι μικρομεσαίε, αποτυγχάνουν και οι επιχειρηματίε. Θα σα πούν ότι έχουν, ε, αν έχουν πετύχει, ότι πρώτα δοκίμασαν 10 φορέ και απέτυχαν και μετά τα κατάφεραν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ανοιχτά διαφανή κεφάλαια, ε, αγορέ κεφαλαίων, ανοιχτέ διαφανεί αγορέ κεφαλαίων που μπορούν να έχουν πρόσβαση οι επιχειρηματίε. Όχι υπάρχουσε, ε, ούτε τα κεφάλαια κινδύνου που έχουν πολύ περιορισμένη και αυστηρή προσέγγιση στα πράγματα τώρα. Εγώ, εσείς, οποιοδήποτε από εμά ε, θα επένδυε στην ε, μικρομεσαία επιχειρήση που θα πίστευε, εάν πίστευε ότι θα μας έφτανε, θα έφερνε ανάπτυξη στην κοινωνία, θα πρόσφερε ωφέλη σε όλους, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης. Καταλαβαίνουμε όλοι τους κινδύνους από μια επένδυση. Ο κόσμος αγοράζει σπίτια, είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής. Μέρος της καθημερινής ζωής. Ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει αποτυχία. Το crowdfunding λοιπόν ε, ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια και μεγάλες διαστάσεις πήρε τα τελευταία 5. Εδώ μιλάμε για 2 δις ευρώ ετησίως για χρηματοδότηση μικρομεσαίων και χωρίς κρατικές βοήθειες, 2 δις ευρώ, 30-40% στήριξη από κυβέρνηση από το EIF, που είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Ευρώπη, με κεφάλαια κινδύνου. Αλλά εδώ μιλάμε για crowdfunding, για, μικρό, για μικρό, μικρές διαστάσεις, για ενώσεις, για μικρομεσαίες, χωρίς κρατική βοήθεια, με μικρούς επενδυτές που δεν θεωρούνται επιχειρηματικοί φορείς, ούτε μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εκεί έχουμε στήριξη και στο επιχειρηματικό κεφάλαιο για πέντε χρόνια ε, το πολύ 5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα, ένα άλλο ίδρυμα θα χρειαζόταν πολύ περισσότερα χρόνια για να επενδύσει αναλόγως. Εδώ λοιπόν αυτό που έχουμε εμεί ω πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα. Μπορούμε πολύ γρήγορα να λάβουμε αποφάσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ε, υποφελούμαστε από τι ειδικέ γνώσει άλλων για πολλέ συναλλαγέ που ήδη έχουν σχεδιαστεί ε, υπάρχει αίσθηση των μικροεπενδυτών ότι μπορούν έτσι να αποταμιεύσουν τα χρήματά τους. Κίνδυνοι υπάρχουν και τους ε, αντιμετωπίζουμε. Θέλουμε δηλαδή να βεβαιωθούμε ότι δεν τους πιάνουμε κορόιδα και χάνουν τα λεφτά τους, αλλά αυτό είναι και μέρος της ε, ζωής. Θα συμβεί όπως έχει συμβεί και σε άλλους τομείς. Έχει ήδη συμβεί στον τραπεζικό τομέα, έχει συμβεί στον τομέα των κεφαλαίων κινδύνων, έχει συμβεί στην πολιτική. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να δώσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν, στους καθημερινούς ανθρώπους, ε, στον δρόμο, στη δουλειά τους, που έχουν ένα μικρό εισόδημα, τη δουλειά τους, τη ζωή τους, να πάρουν αποφάσεις και να μπορούν να δράσουν εδώ. Αυτά θα πρέπει να καλύψουμε τους κανονισμούς μας. Δηλαδή να προωθήσουμε τη δράση των μικρών επενδυτών, με το τραπεζικό σύστημα με άλλο τρόπο. Αλλά έτσι θα κινητοποιήσουμε το κεφάλαιο που αυτή τη στιγμή έχει μείνει στου λογαριασμού τη τράπεζα, του αποταμιευτικού. Έτσι θα επενδύσουν οι πολίτε στην πραγματική οικονομία. Εάν φαντάζεστε ότι το Α.Ε.Φ. το κόσμο θα κάνουν την δουλειά που θέλουμε δεν θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή μπορεί κάποιος που μόλις ξεκίνησε να υποβάλει αίτηση και να πάρει πολύ γρήγορα τα χρήματα που χρειάζεται, όχι. Με αυτά τα προγράμματα δεν αρκεί. Το crowdfunding αυτή τη στιγμή είναι μια μικρή αγορά με επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν τον κίνδυνο να φτιάξουν αυτές τις πλατφόρμες. Λειτουργεί σαν αγορά όπου οι πολιτές και οι αγοραστές ε, συναντώνται και όλα αυτά πρέπει να λάβουν επισημότερη μορφή. Για την ώρα έχουμε συνεργασία με πρόσωπους από χρηματιστήρια, επιχειρήσεις, τράπεζες, ε, από τα κεφάλαια κινδύνου. Αυτοί θα πρέπει όσα αναπτύσσουμε να τα δουν ως ευκαιρίες. Να μας δώσουν την κατάλληλη διάρθρωση, δομή και τα πλεονεκτήματα στην ενημέρωση, ώστε να μπορέσουμε να ωφελήσουμε τους μικρούς επιχειρηματίες. Σκεφτείτε τώρα, 10.000 δάνειο σε μια μικρομεσαία. Ποια τράπεζα θα το κάνει σήμερα. Σκεφτείτε τι δουλειά χρειάζεται μια τέτοια τράπεζα. Αν όλα αυτά γίνουν μέσω υπολογιστή, αν μπορεί αυτή η διαδικασία να επιταχυνθεί, τότε θα γίνουμε πολύ αποτελεσματικότεροι στην ε, εκδαμείευση κονδυλίων. Και θα μπορέσουμε να χρηματοδοτούμε ρηγορότερα τι μικρομεσαίε. Για μένα λοιπόν αυτό είναι ζωτική σημασία και δεν νομίζω ότι η συζήτηση που πρέπει να κάνουμε είναι εάν θέλουμε να γίνει αυτό ή όχι, αν το επιτρέψετε ή όχι, πρέπει να σκεφτούμε πώς η ψηφιακή επανάσταση αλλάζει την ζωή μας και πώς οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι ίσως μια από τις τελευταίες πτυχές όπου μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά πάτε στην αγορά της Λιανικής και ζητήσετε να μάθετε τι ε, αλλαγή έχει, κάνει, έχει φέρει το Amazon και το eBay, έχει καταστρέψει κάποιες μεγάλες εταιρείες ε, το Amazon και το eBay. Ε, δείτε λοιπόν και σε ανάλογους τομείς τι συμβαίνει. Ε, αυτή τη στιγμή οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μπορούν να εκτελούνται μέσω υπολογιστή και το crowdfunding είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Σας ενθαρρύνω λοιπόν να σκεφτείτε διαφορετικά την ανάληψη κινδύνου, το ρόλο των πολιτών και αν σκεφτείτε σκέφτεστε την πρόσβαση στην αγορά, μην σκεφτείτε μόνο τα κεφάλαια κινδύνου, μην σκεφτείτε τα επιχειρηματικά κεφάλαια μόνο, αλλά ένα οικοσύστημα που όλα αυτά συλλειτουργούν. Με φορολογικά κίνητρα για του επενδυτέ, ώστε όταν αναλαμβάνουν ένα κίνδυνο και επενδύουν σε μια μικρή επιχείρηση να ξέρουν ότι μπορεί να αποτύχουν και αν αποτύχουν να μην τιμωρηθούν γι' αυτό, αλλά να έχουν ε, κάποιο κέρδο, ε, κάποια επιστροφή. Διότι μπορεί να ε, επενδύσουν σε 10 εταιρείε και οι 5 να πτωχεύσουν. Θα τα χάσουν αυτά τα λεφτά. Οπότε καλό θα είναι τουλάχιστον να έχουν κάποιο κέρδο από τα υπόλοιπα. Να καταλάβετε λοιπόν ότι χρειάζεται εδώ και καλλιέργεια, μόρφωση. Δηλαδή ξεκινάει αυτού του είδου η καλλιέργεια νοοτροπία από την ηλικία των τριών για να μάθει κανεί την επιχειρηματικότητα και την χρηματοδότηση. Ε, εάν ξέρατε τι συμβαίνει στην ε, κοινωνία γενικότερα, 40 με 45% των συμπολιτών μας δεν μπορούν να υπολογίσουν τι γίνεται με τα επιτόκια. Πώς να επιβιώσουν αυτοί. Χρειαζόμαστε μια νέα γενιά επιχειρηματιών και αυτό πρέπει να ξεκινήσει πολύ νωρίς. Και επίσης να σκεφτούμε και τη δουλειά των κυβερνήσεων στην απόδοση των κονδυλίων. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι κινητήριο δύναμη οι κυβερνήσει όπω είπατε εσεί. Λένε ότι έχουν στρατηγικέ συγχρηματοδοτήσεων οι κυβερνήσει. Εάν δεν βρεθούν επενδυτέ, πώ θα λειτουργήσουν οι αγορέ. Εκεί πρέπει να πάρει κανεί ε, πρωτοβουλία και να αναλάβει δράση για να χρηματοδοτήσει. Χρηματοδότηση λοιπόν από φορέ τη κυβέρνηση ήδη υπάρχει, αλλά απόδοση κονδυλίων μέσω του crowdfunding είναι ένα τρόπο για να φτάσουν αυτά τα κονδύλια επιτέλου στι μικρομεσαίε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ήρθαμε κοντά στην πραγματική ζωή με τις παρουσιάσεις και τις ομιλίε σας. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Ντεμπάκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους δύο μιλητές, τους γνωρίζω πολύ καλά. Μίλησαν για την λογική ανάληψη ρίσκου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι καινοτόμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα δρουν στο περιβάλλον που πραγματικά τους αξίζει. Ακούω και την έκκλησή σας για την αφύπνιση των ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι πολύ σημαντικό στο Κοινοβούλιο να συζητούμε τι κάνουμε με το δημόσιο χρήμα, το οποίο λειτουργεί ως μοχλός, ως ένα αρκτήριο λάκτισμα, όμως τα ιδιωτικά κονδύλια είναι αυτά που θα χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη των μελλοντικών επιχειρήσεων και συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Έχω όμως δύο-τρεις ερωτήσεις να σας υποβάλω. Κάτι το οποίο με απασχολεί στη συζήτηση με τους επιχειρηματίες είναι το εξής. Ότι εμάς μας χρηματοδοτεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα βεβαίως στην Ευρώπη, οι τράπεζες οι ίδιοι επιχειρηματίες δεν είναι ανοιχτοί, δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχουν και εναλλακτικέ λύσεις και διαφορετικές λύσεις. Χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας, μια αλλαγή αντιλήψεων, όχι βεβαίως να αντικατασταθεί ο, ο τραπεζικός δανεισμός, αλλά να υπάρξει και ε, επένδυση με ίδια ε, κεφάλαια και κεφάλαια που συγκεντρώνονται από την αγορά. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, μιλήσατε για την καθαρή τεχνολογία, για την πράσινη ανάπτυξη. Υπάρχει αγορά για αυτές τις επιχειρήσεις, το επενδυτικό του σχέδιο είναι στέρεο, αξίζει όλο και περισσότερα κεφάλαια να ε, ενδιαφερθούν για αυτό το τομέα. Τι πιστεύετε Ισχύει αυτό για την καθαρή τεχνολογία και για τις ε, ε, εταιρείε που ασχολούνται με την πράσινη ανάπτυξη. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προσελκύσουμε πολύ περισσότερα κεφάλαια ε, σε αυτό το τομέα. Και τέλος, για το crowdfunding. Δεν είναι εργαλείο ιδίων κεφαλαίων. Δεν μπορούν να έχουν απόδοση αυτοί που επενδύουν, όπως γίνεται με τα επενδυτικά κεφάλαια που είναι με σύμπραξη. Ισχύει αυτό. Εταιρείε στην καθαρή τεχνολογία, στις ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια έχουν, ε, επιτύχει, έχουν επιτύχει πολλά και μπόρεσαν να δώσουν μια κάποια απόδοση στους αρχικούς επενδυτές. Έτσι έχω ακούσει. Ποια είναι η γνώμη σας. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ο κύριος Πολ Ρούλικ, ο σκιώδη εισηγητή. παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η παρεμβάσεις δείχνουν πολύ καλά προς τα που θα πρέπει να κινηθούμε στην Επιτροπή ε, Προπολογισμού. Παρουσίασα μια πρόταση για τις ε, γυναίκες ε, επιχειρηματίες. Μπορείτε να μας πείτε παραδείγματα για το πώς το Business Angels στο τομέα του crowdfunding μπορούν να δραστηριοποιηθούν. Χρειαζόμαστε λοιπόν βέλτιστες πρακτικές, παραδείγματα, benchmarks στον τομέα αυτό, αλλά αυτό δεν γίνεται χωρίς κάποιες ηγετικές φυσιογνωμίες που θα μας δείξουν πώς τα πράγματα θα διαμορφωθούν στην πραγματικότητα. Υπάρχουν κάποια καλά παραδείγματα και θα πρέπει να τακμηριωθούν, να δοθούν κίνητρα προκειμένου κάποιος να βγει στη δημοσιότητα και να πει ότι ναι, ξέρω πώς πάει, ξέρω πώς λειτουργεί αυτή η κατάσταση, έχω μάθει τα μέσα που χρειάζονται και είμαι εδώ διατεθειμένος να σας δείξω ένα μικρό ατμήμα. Αλλά αισθάνομαι ευθύνη για την διαφάνεια και θέλω να υπάρχει πρακτική καθοδήγηση και από την κοινή γνώμη για να αποδείξουμε ότι πρόκειται για ε, έντιμα, ειλικρινά προϊόντα που αποδίδουν. Θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε πώς ε, σε αναλήψης κινδύνου, πώς θα υπάρξει ένα ε, πριν κινδύνου. Να υπάρχει λοιπόν μια κουλτούρα κινήτρων. Τι κίνητρα μπορούμε να δώσουμε για να ενθαρρύνουμε. Γιατί ξοδεύει ο κόσμος χρήματα στο λότο και στο τότο και στα υπόλοιπα και στους ε, λαχιοφόρους αγορές όπου ποτέ δεν κερδίζει χρήματα. Είναι μάλλον πολύ μικρή απόδοση και όχι εδώ. Και τελικά μόνο ο ιδιοκτήτης λοταρίας είναι αυτός που επωφελείται. Χρειάζεται ίσως και διαφημίσεις ε, για πολλά προϊόντα πληρώνουμε ένα 30% παραπάνω για τα ποσά αυτά. Δεν θα είχε νόημα να εστιαστούμε στις μικρομεσαίες αυτές τις επιχειρήσεις και να δούμε τι γίνεται σε ό,τι αφορά την ε, προπολογισμό ακόμα και του Ιούνκερ και την απόδοσή του. Σας ευχαριστώ πολύ. Το ευχαριστούμε τους συζητές μας. Πολλές ερωτήσεις ακούσαμε. Και για τους προηγούμενους ομιλητές. Απάντησαν λοιπόν ε, οι πρώτες ομιλητρίες. Έχει έρθει η ώρα να απαντήσετε κι εσείς. Α, έχουμε κι άλλη μια ερώτηση. Έχετε το λόγο. Πάρα αυτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια ερώτηση λίγο συμπληρωματική. Επερώτηση. Αφού ευχαριστήσω για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις. Εδώ μιλάμε πάντοτε για χρηματοδότηση χρηματοδότηση των μικρομεσαίων που έχουν κάτι να παράγουν για να πάει στην αγορά. Είτε ένα νέο προϊόν, είτε τέλο πάντων κάτι που είναι αντικείμενο εμπορία. Ξέρουμε σήμερα ότι ο κυκλός ζωή των προϊόντων όλο ένα και περιορίζεται. Οι επιχειρήσεις που θέλουν να είναι βιώσιμες, να έχουν μια δράση μακροπρόθεσμη, πρέπει συνεχώς να καινοτομούν Όποιος λοιπόν έχει ήδη εμπορευτεί ένα προϊόν θα πρέπει να αναζητήσει το επόμενο υπολογίζοντας το, τέλος κύκλου ζωής του ε, προϊόντος. Για την κοιλάδα του θανάτου της καινοτομία λοιπόν τα πράγματα είναι πολύ περίπλοκα για τις μεγάλες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλα αυτά τα επιχειρηματικά κεφάλαια, τα κεφάλαια κινδύνου, τα crowdfunding με έναν πυλώνα που πιστεύω ότι πρέπει να είναι δημόσιο, ένα ταμείο για την καινοτομία ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν απευθεία σύνδεση με τα κέντρα γνώσης. Δηλαδή, Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί γύρω από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θα πρέπει να διαρθρώνονται σε ένα κεντρικό σκελετό, ο οποίος να στηρίζει την κοινοτομία και να φροντίζει για τα διπλώματα τεχνίας. Θα ήταν πιο πλήρες έτσι το σύστημα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και να συμπληρώσω τα προηγούμενα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω κάτι πιο ε, ευρύ για τα ιδιωτικά και δημόσια κονδύλια στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, ενδεχομένως μπορείτε εσείς να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχετε το λόγο. Ναι. Πολλές ερωτήσεις μου έχουν τεθεί. Καταρχάς να επιβεβαιώσω κάτι που έχω ακούσει. Πράγματι, πέρα από τη χρηματοδότηση των ε, τραπεζών υπάρχουν και άλλα μέσα χρηματοδοτικά, τα συζητήσαμε και υπάρχουν και έχουν μεγάλη αξία. Έχουμε το venture capital, έχουμε τους επιχειρηματικούς αγγέλους, το business angels. Είναι σαν να ε, κάνουμε έγχυση βακτηρίων σε έναν μικρό οργανισμό, σε έναν ζώντα μάλλον οργανισμό, έτσι ώστε να ξυπνήσει, να μην είναι σε χειμερή ανάρκη. Μπορεί ενδεχομένω να έχει κάποιες εξάψεις, μία μικρή άνοδο πυρετού, αλλά έτσι θα καταπολεμήσει τα προβλήματα και θα ε, γίνει καλά. Τώρα για το θέμα των ε, καθαρών τεχνολογιών και όλης αυτής της βιομηχανίας. Δεν είμαι ειδικό. Είναι όμως μια βιομηχανία η οποία λειτουργεί με απελπιστικό τρόπο θα έλεγα γιατί είναι υψηλής εντάσεως κεφαλαίου χρειάζεται πάρα πολλά ιδιωτικά κεφάλαια και συμπληρωματικά χρειάζεται και δημόσια κεφάλαια για να ε, υλοποιηθεί και να γίνουν οι σωστές ε, τεχνολογικές και επιχειρηματικές επιλογές. Είναι μια νέα βιομηχανία, ένας νέος κλάδος. Το επιχειρηματικό μοντέλο δεν έχει ξεκαθαρίσει. Δεν είναι πολύ σαφές πόσοι οι επενδυτές θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους, θα έχουν κάποια απόδοση. Τώρα, ως προς τα, τους ρόλους πρότυπα, είναι πολύ σημαντική και σε βελγικό επίπεδο και αλλού. Ε, το VCA, το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, Business Angels, ε, και στις γειτονικές χώρες δίνεται, διαχέεται, διαδίδεται το παράδειγμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πώς μπορεί κανείς να έχει μια θετική αφήγηση ακόμα και αν προσπαθεί το, να βρει το δρόμο του μέσα σε ένα ναρκοπαίδιο. Και το πιο σημαντικό, και το λέω αυτό υπέρ του crowdfunding βέβαια, είναι το εξής. Εμείς δεν έχουμε εισιτήρια των 300 ευρώ, έχουμε εισιτήρια τουλάχιστον μισού εκατομμυρίου ευρώ για τους επενδυτές. Στοχεύουμε σε ακριβώς αυτούς τους επιχειρηματίες, αυτούς που τα κατάφεραν πριν αυτοί που επενδύουν σε εμά δεν είναι το παλιό χρήμα εντό εισαγωγικών, είναι το καινούριο χρήμα. Είναι επιχειρηματίες που καταλαβαίνουν την προσέγγισή μας και θέλουν να βάλουν χρήματα πάνω στο τραπέζι. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε φυσιολογικά πλαίσια ε, παρετούνται εν, μέρο, μέρη από κάποιες από τις ανέσεις τους, στη ζώνη άνεσής τους, σε μέσα σε αυτό το δακτύλιο που ε, διαβιούν, προκειμένου ε, να συμμετάσχουν σε κάτι πιο σημαντικό, σε κάτι ενδεχομένω ε, κερδοφόρο. Είναι σημαντικά δηλαδή τα κίνητρα. Τα κίνητρα τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να έχουμε πλατφόρμες συνεπενδύσεων. Να συμπληρώσουμε όλα αυτά τα έργα με δημόσιο χρήμα και έτσι μπαίνουμε σε έναν πιο ενάρωτο κύκλο, πιο πιθανό ε, να πετύχουμε ε, και να έχουμε επιτυχία. Δεν θα πρέπει ναι είναι υποκατάσταση, να έρχεται το ιδιωτικό χρήμα να υποκαταστήσει το δημόσιο, ούτε αντιστρόφως βεβαίως. Σίγουρα οι εταιρείε ακολουθούν ένα συγκεκριμένο κύκλο ζωής. Η βιομηχανία μας το καταλαβαίνει αυτό πάρα πολύ καλά. Οι συνάδελφοι βλέπουν τις πιο όριμες εταιρείε. Εάν η επιχείρησή σας ε, αναπτύσσετε και είναι πολύ επιτυχημένη, κάποια στιγμή θα φτάσετε στο μέγιστο επίπεδο και μετά από αυτό θα φθείρει η εταιρεία αυτή, θα φθαρεί. Και αυτό οφείλεται ε, στις πολύ γρήγορες τεχνολογικές καινοτομίες που θα υπάρξουν. Οι επιστήμες της ζωής, τα νέα φάρμακα, οι νέες θεραπείες, η νέα τεχνολογία. Ε, δεν μπορούν να υπάρχουν ακολουθώντας τι πεπατημένοι. Χρειαζόμαστε λοιπόν τους επιχειρηματικούς αγγέλους, τα venture capital, ακριβώς για να ε, έρθουν και να συμβάλλουν όταν οι εταιρείε έχουν φτάσει στο απόγειό τους και είναι έτοιμες πλέον να πάρουν την κατηφόρα. Ξέρετε, Πολύ συχνά οι αλλαγές δεν είναι ευπρόσδεκτες. Κάθε αλλαγή δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα και υπάρχουν νεύρα, υπάρχει ένταση, υπάρχει εκνευρισμός. Νομίζω ότι αυτά είναι που πρέπει να ξεπεραστούν και έτσι θα έχουμε καινοτομία και θα μπορέσουμε να, και να δημιουργήσουμε και να στηρίξουμε ε, τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Για να απαντήσω στις ερωτήσεις σε ό,τι αφορά την ε, συνειδητοποίηση για τα μέτρα για το επιχειρηματικό κεφάλαιο. Νομίζω ότι πολλά έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την ε, τράπεζα. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε χρόνο υπάρχουν νέοι απόφοιτοι και αν δεν έχουν ακολουθήσει τις σχετικές ε, σπουδές δεν ξέρουν τι είναι το venture capital, το κεφάλαιο κινδύνου και επειδή ε, πολλοί επιχειρηματίες δεν έχουν σπουδάσει οικονομικά, δεν ξέρουν απαραίτητα τι είναι το κεφάλαιο κινδύνου, γιατί δεν διδάσκονται απαραίτητα τα πράγματα αυτά στο σχολείο, δεν ξέρουμε απαραίτητα τι είναι αυτό το επιχειρηματικό κεφάλαιο. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε με το χρέο και πώ θα το αντιμετωπίζουμε. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε και εδώ θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη βάρος. Ε, επιστροφή στο crowdfunding. Ναι, φυσικά και υπάρχει τέτοια ε, απόδοση του crowdfunding, συγγνώμη. Υπάρχει μια βάση δωρεών όπου θέλουμε να δούμε επιτυχία και αυτό είναι μεγάλο κίνητρο. Υπάρχει λοιπόν και μία εκστρατεία ανταπόδοσης όπου υπάρχει ε, απόδοση σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις για τη δημιουργία ε, προσόδων. Υπάρχει ένα προϊόν. Αυτό εξαρτάται από το κίνητρο τη χρηματοδότηση. Δεν πρόκειται για επένδυση, πρόκειται για χρηματοδότηση, όπου δίδεται χρήματα για κάποιον για να προωθήσει μια ιδέα. Και υπάρχει και το crowdfunding για το επιχειρηματικό κεφάλαιο, όπου γίνεται λοιπόν επένδυση με επιχειρηματικό κεφάλαιο. Αν οι επιχειρήσεις λοιπόν δείξουν, ε, έχουν επιτυχία, υπάρχει απόδοση. Το θέμα είναι κατά πόσο θα υπάρχει επιτυχία και κατά πόσο θα υπάρχει καθοδήγηση προκειμένου να πετύχουν και θα πρέπει ο επενδυτής να κατανοήσει ότι είναι πιθανό να μην υπάρχει η ανάπτυξη που περιμένει ή να μην υπάρχει η σωστή επιτυχία, άρα προσοχή στις επενδύσεις. Και αυτό έχει να κάνει με τα θέματα ευαισθητοποίησης που τονίσαμε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους ε, ιδιώτες. Ο δανεισμός δουλεύει πάρα πολύ καλά στο crowdfunding και σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πολλά τέτοια έργα χρηματοδοτούνται. Είναι λοιπόν μια λύση για πολλά ζητήματα, για τα πάντα. Για την πόλη του, το Δήμο του Παρισίου, για παράδειγμα, που έχει χρησιμοποιήσει crowdfunding, μπορεί λοιπόν να ε, υπάρξει απόδοση. τα business angels δεν είναι απαραίτητα πάρα πολύ ανοιχτά. Δεν μιλούν δημόσια για το τι κάνουν, αλλά τα επόμενα εβδομάδα θα γίνει μια διάσκεψη στο Παρίσι και θα υπάρχει και η πρόεδρος του Business Angels Network και των Ευρωπαϊκών Σχετικών Δικτύων που θα μιλήσουν γιατί κατανοούν ότι είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να συνεργαστούμε. Και υπάρχουν και διάφορες οργανώσεις και των ε, μετόχων και διαφόρων οργανισμών. Δεν υπάρχει να έρθει κάποιο ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώ. Για να δοθούν κίνητρα λοιπόν για τους μικρούς επενδυτέ. Νομίζω ότι τα κίνητρα έχουν να κάνουν ε, με την ελπίδα οικονομικής απόδοσης ε, και η επιθυμία να αλλάξει ένα μικρό κομμάτι του κόσμου. Αυτό ισχύει και για τα κεφάλαια κινδύνου δεν είναι πάντα το θέμα η οικονομική απόδοση και θα πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος αυτή την ιδέα ότι κάθε απόφαση, ακόμα και στις αγορές αποφάσεων, γίνεται μόνο για οικονομικούς λόγους. Ίσως σε κάποιους τομείς ε, συναλλαγών, αλλά πάντα υπάρχει και η διάσταση του συναισθήματος, του ανθρώπινου συναισθήματος. Mm. Το κύκλος ζωής του προϊόντος αποτελεί ένα θέμα ασφαλώς. Δεν έχω την απάντηση να σας δώσω αν θέλετε να χρηματοδοτηθεί μια επιχείρηση μέσω της τράπεζα, υπάρχει μια διαδικασία, πρέπει κανεί να πάει στην τράπεζα να ζητήσει την, ε, το δάνειο. Παίρνει πολύ χρόνο, παίρνει πολύ ενέργεια. Το ίδιο ισχύει και για τα κεφάλαια κινδύνου, αν χρειάζεται χρηματοδότηση κάθε δύο χρόνια. Και το ίδιο ισχύει και με το crowdfunding. Είναι χρονοβόρο, είναι κοστοβόρο, πρέπει να υπάρχει μια εκστρατεία, να οικοδομηθεί ένα δίκτυο να ψάξει κανείς πλατφόρμες crowdfunding σε διάφορες περιστάσεις κατά τη διάρκεια των ετών προτού φτάσει σε ένα καλό επίπεδο επένδυσης, αλλά αποτελεί μια ευκαιρία για μικρά ποσά με μια περιορισμένη προσπάθεια κάθε χρόνο και αυτό για να χρηματοδοτηθούν και καινοτομίε νέων προϊόντων. Το πρόβλημα είναι, σε ό,τι αφορά τις ε, χρηματοδοτήσεις γρήγορες, δεν μπορεί να επιληθεί. το κοινό μπορεί να υποστηρίξει κάποια μέσα και οι κυβερνήσεις μπορούν να υποστηρίξουν τέτοια, τέτοια μέσα. Στη Βρετανία 30 δισεκατομμύρια λίρες για την ε, α, χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω crowdfunding. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία και ορίστηκαν στους επενδυτές ε, που επένδυσαν μέσω της πλατφόρμας. Πρόκειται για μια καλή ιδέα. Η αγορά λοιπόν αποφασίζει ποιες επιχειρήσεις θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν και συγχρηματοδοτική κυβέρνηση είναι καλή ιδέα. αυτό είναι ο ρόλος των ε, μέσων αυτών. Θέματα IP, ε, πνευματικής ιδιοκτησίας, υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν είναι κάθε επιχείρηση διατεθειμένη να ζητήσει χρηματοδότηση crowdfunding, γιατί είναι πολύ δημόσιο χαρακτήρα Θα πρέπει να δημοσιεύσει το τι κάνει, κάποιε συγκεκριμένε πληροφορίε. Οι πιο πολλοί που κάνουν και χρησιμοποιούν το crowdfunding δεν πρόκειται να σα κλέψουν την ιδέα σα, αλλά φυσικά υπάρχουν και ανταγωνιστικέ επιχειρήσει. Από την άλλη, κοιτώντα την πραγματική καινοτομία που έχει επηρεάσει την, την κοινωνία μα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, πάντα τα προϊόντα αυτά δεν είχαν προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτός που έφτιαξε τον τροχόν δεν είχε ε, προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτός που ε, δημιούργησε τον γραπτό λόγο δεν είχε πνευματική προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα. Άρα ίσως κάποια πράγματα δεν θα έπρεπε να είναι προστατευμένα και κοιτώντα και την επιτυχία του λογισμικού ε, open source ανοιχτή πηγή, προς την κατεύθυνση αυτή κινείται. Ότι μπορεί κανείς παρόλα αυτά να οικοδομήσει κάτι πολύ χρήσιμο και να αποφελήσει την, οικογένεια, την κοινωνία μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις και τις ε, ε, ομιλίες σας, αλλά επειδή ε, έχω λάβει και την υποχρέωση να συντάξω ένα κείμενο με τα συμπεράσματα από τη συνάντηση 28 επιτρόπων και 22 προέδρων κοινοβουλευτικών επιτροπών θα ήθελα να ζητήσω από τον ε, πρώτο αντιπρόεδρο, συμπρόεδρο για τη σημερινή ε, συνεδρίαση, δηλαδή την κυρία Πατρίτσια Τόγια, να αναλάβει την Προεδρία για το τρίτο σκέλος της ε, ακροασής μας. Παρακαλώ. Ωραία, συνεχίζουμε αυτή την ενδιαφέρουσα ακρόαση. Περνάμε στο τρίτο πάνελ. Μετά από όλα τα τόσο σημαντικά θέματα, περισσότερο οικονομικά που ακούσαμε, ας δούμε πώς μπορούμε να ε, προωθήσουμε το δυναμικό με μια καινοτόμα προσέγγιση για τις καινοτόμες μικρομεσαίες. Δηλαδή αναζητούμε νέους δρόμους και νέα βήματα σε αυτήν την πορεία της ευρωπαϊκής ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή οικονομία. Πρώτη παρέμβαση, ο κύριος Ζωάου Βασκονσέλος, τελεστικός διευθυντής της Startup Lisboa για τις νεοφιλείς επιχειρήσεις της Πορτογαλίας. Για 10 λεπτά, παρακαλώ. Good morning. Thank you, uh, Chairman, uh, Καλημέρα σας ε, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η Startup Lisboa είναι μια ιδιωτική ένωση με κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βασικό στόχο τη στήριξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων, των νεαρών επιχειρήσεων στην πόλη της Λισαβόνας. Ε, ήδη λειτουργούμε εδώ και τρία χρόνια και είμαστε μέρος όπου δίνουμε ε, επενδύσεις ε, και επιτρέπουμε στους επενδυτές επίσης να λάβουν ενημέρωση. Σε ένα παλιό κτίριο στο ιστορικό κέντρο της Λισαβόνας έχουμε δραστηριότητες από mentoring μέχρι ενημέρωση. Έχουμε έναν ειδικό χώρο για την ε, εκπαίδευση και φροντίζουμε αυτή η γνώση που προσφέρουμε να μεταφραστεί σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Ουσιαστικά δηλαδή ο στόχος είναι να βρούμε επενδυτές ή και πελάτες για νεοσύστατες επιχειρήσεις. Όπως ε, σας είπα ξεκινήσαμε το Φεβρουάριο του 2012 την δράση μας και εκτοτέ έχουμε εξετάσει 3.000 υποψηφιότητες από όλο τον κόσμο. Έχουμε 28, ε, ε, συμμετοχές από 28 εθνικότητες και ε, οι υποψηφιότητες που εξετάσαμε και εγκρίναμε έφτασαν τις 190-200 επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή 70 επιχειρήσεις στηρίζονται και το μέσο χρονικό διάστημα που μένουν κοντά μα οι εταιρείε είναι περίπου ένας χρόνος. Οι επιχειρήσεις που εξετάσαμε πριν από τρία χρόνια ήταν κυρίω από το χώρο της ψηφιακή οικονομίας, του διαδικτύου, του κινητού διαδικτύου, του διαδικτύου στα κινητά δηλαδή και στους υπολογιστές από πέρσι με το νέο μας κτίριο ε, εφαρμόσαμε την ίδια ε, αρχή με, τις, με τουριστικές επιχειρήσεις, με εμπορικές επιχειρήσεις και ε, έπειτα θα υπάρξει και ένας νέος κλάδος με νέες εταιρείε με, που, θα, που θα τους ζητηθούν αίθουσες, αίθουσες γραφικής στήριξης στην Λισαβόνα πάλι έχουμε 600, 650 θέσεις εργασίας στην Λισαβόνα. Ε, ένα ρεκόρ για, το, για την οικονομική κρίση που γνώρισε η χώρα μας τον τελευταίο χρόνο. Έχουμε περίπου 70 ε, υπευθύνους για mentoring οι οποίοι στην ουσία είναι ιδρυτές επιχειρήσεων. Εκείνοι φέρουν τις εταιρείες στο Startup Lisboa και εκείνοι μετά παρακολουθούν και την εξέλιξή τους. Πολλές φορές μέχρι να βρουν τους πρώτους τους επενδυτές ή τους πρώτους τους πελάτες. Έτσι έχουμε ιδρυτές, γενικούς διευθυντές, γνώστες του θέματος και ευτυχώς ο επιχειρηματικός κόσμος και επιχειρηματικότητα έγινε προτεραιότητα για την Πορτογαλία. Πολύ εντυπωσιακό αυτό σε καιρό κρίσης και λόγω του υψηλότατου ποσοστού της ανεργίας των νέων. Χρειαστήκαμε λοιπόν στήριξη από τις μεγάλες επιχειρήσεις της Πορτογαλίας και είχαμε στήριξη και από την κυβέρνηση και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μεγαλύτεροι υποστηρικτέ λοιπόν του Startup Lisboa είναι ο Δήμος τη Λισαβόνας με ε, μια τράπεζα που έχει προσφέρει τη στέγαση της ε, Startup Lisboa και συνειδητές όχι νομικός ε, αλλά ατύπως είναι 30 επιχειρήσεις η Microsoft η Price και άλλες και για τους επενδυτές είπαμε 28 εθνικότητες και εταιρείες που λειτουργούν σε 30 διαφορετικές αγορές. Η Startup Λισμπόα αποδεικνύει κάτι που νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει παντού, όχι μόνο στην Πορτογαλία. Κάτι που αποδεικνύει την δύναμη του οικοσυστήματος, όπως έλεγα. Οι επιχειρήσεις δεν αναπτύσσονται ε, στον τομέα τουλάχιστον που γνωρίζουμε δεν στηρίζονται μόνο από τα κεφάλαια για την καινοτομία, αλλά αναπτύσσονται μέσω των πελατών και των επενδυτών τους. Το ε, Silicon Valley ε, λόγου χάρη. Ε, πολλές είναι εταιρείε που ιδρύονται στην Βοστόνη και παρόλα αυτά φτάνουν στο Silicon Valley. Στην Ευρώπη λοιπόν επενδύουμε στην επιστήμη, την κοινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη, στα πανεπιστημιακά κέντρα. Τώρα Πρέπει να περάσουμε σε μια νέα φάση επιτέλους. Πρέπει να επενδύσουμε και να αναζητήσουμε ανάλογους πόρους για να βρούμε πελατολόγιο στις εταιρείες Η επιστήμη και γνώσεις αυτές να μεταφραστούν σε προϊόντα, σε πλούτο και σε θέσεις εργασίας. Στην Πορτογαλία τα πανεπιστήμια δεν είναι πηγή για τον επιχειρηματικό κόσμο. Τα τεχνικά ιδρύματα ιδίω, διότι σήμερα τα περισσότερα μαθήματα αυτά που διδάσκονται, οι κύκλοι μαθημάτων, καλύπτονται στις θέσεις εργασίας τους και στην αγορά εργασίας και από την κεντρική και από την ανατολική Ευρώπη πολλές φορές. Όμως, στους ε, μηχανικούς λόγω χάρη στα πολυτεχνία, ε, ε, οι νέοι συνήθως παίρνουν ε, καλύτερη μόρφωση από τη γενιά των γονιών τους. Αλλά είναι πολύ δύσκολο επίσης να πείσει έναν νέο να γίνει επιχειρηματίας, να ιδρύσει τη δική του εταιρεία. Όμως όταν κανείς θα αποφασίσει θα προχωρήσει. Και εκεί είναι που παραμένουμε εμεί. Οι περισσότεροι επιχειρηματίε με του οποίου ασχολούμαστε είναι νέοι, κατά μέσο όρο 28 ετών, με ήδη κάποια επαγγελματική κατάρτιση. Ε, η μεγαλύτερη πηγή που μα τροφοδοτεί είναι οι μεγάλε εταιρείε, οι Goldman Sachs, άλλε μεγάλε τράπεζε, η Microsoft. Και οι νέοι αυτοί ουσιαστικά θέλουν να ιδρύσουν μια δική του εταιρεία. Τι περισσότερε φορέ Οι νέοι αυτοί πρέπει να ξέρουν ότι μπορεί να αποτύχουν, ότι μπορεί να μην λειτουργήσει η ιδέα τους, να μην δώσει αποτελέσματα και σε κάθε περίπτωση τα πανεπιστήμια της Πορτογαλίας πάντα ήταν μεγάλοι ε, ε, συνομιλητές του επιχειρηματικού κόσμου. Όλοι ήξεραν ότι αν θέλουν να περάσουν στον κόσμο των επιχειρήσεων έπρεπε να περάσουν από τα πανεπιστήμια. Όμως αυτό τελικά δεν έχει φέρει αρκετό κέρδος. Τώρα η Startup Lisboa που έχει συνεργασία με πολλές εταιρείε βλέπει ότι μπορεί να αλλάξει η τάση αυτή. Δηλαδή το πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ καλό για το σχεδιασμό του προϊόντος, πολύ καλό ακαδημαϊκά και θεωρητικά, αλλά δεν φτάνει για να ιδρύσει κανείς μια επιχείρηση. Πρέπει να βρει κανείς που θα λειτουργήσει, να ιδρύσει την εταιρεία, χρειάζεται πείρα από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Αυτά δεν διδάσκονται στους κύκλους ε, των μαθημάτων και στο, στο επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε οικοσυστήματα όπως έκανε η Λισαβόνα. Βλέπουμε ε, η Λισαβόνα να έχει λάβει ε, βραβείο για το 2015 ε, από την Επιτροπή των Περιφερειών ως χώρος δημιουργίας επιχειρηματικότητας. Εδώ μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε ε, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους οικονομικούς κλάδους και να απευθυνθούμε σε πολλές κατηγορίες επενδυτών. Είδαμε ότι για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι καθοριστικός ο ρόλος των τοπικών κυβερνήσεων και των ε, ε, δημοτικών αρχών. Υπάρχει και ένας ανταγωνισμός μεταξύ αστικών κέντρων, δηλαδή βλέπουμε να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ χωρών όπως, όπως το Βερολίνο ή η Βοστόνη, το Λονδίνο και το Παρίσι. Εδώ μπορούν να παίξουν ένα ρόλο και οι δημοτικές αρχές. Μπορούν να δώσουν κίνητρα, να ε, καλέσουν σε συμμετοχή τις μεγάλες εταιρείες, οι τεχνολογικές νεοσύστατες εταιρείες δεν είναι μόνο μία πηγή που τροφοδοτεί τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά είναι μια πηγή καινοτομία. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να ανακαλύψουν ότι είναι πολύ φτηνότερη, πολύ αποτελεσματικότερη, πολύ ευφιέστερη η επιχειρηματικότητα που έρχεται από νοσίστες εταιρείες από ό,τι από άλλες ε, κλασικές πηγές. είδαμε μια εταιρεία να φτάνει στο Silicon Valley ξεκινώντας από το startup Λισμπόα. Βλέπουμε λοιπόν πώς μπορεί να εξελιχθεί μια επιχείρηση που αρχικά δεν μπορεί κανείς να προβλέψει την πορεία της. Επίσης, η επιχειρηματικότητα δεν είναι μια μαγική ιδιότητα κάποιου που αποφασίζει ξαφνικά να εφαρμόσει επιχειρηματικούς στόχους. Χρειάζονται πολλές ιδέες και πολλά στοιχεία για να πετύχει κανείς στον κόσμο των επιχειρήσεων. Οι εταιρείε λοιπόν θα πρέπει να ε, επενδύουν στις νεοσύστατες και όσοι επιχειρούν να γνωρίζουν ότι μετά την επιτυχία τους πρέπει να ε, συνεχίσουν την προσπάθεια. Εδώ μιλάμε για την πρώτη γενιά νέων Πορτογάλων επιχειρηματιών. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μπορεί να έχουν πολλά προσόντα ως πολύ περισσότερα προσόντα από τους ανταγωνιστές τους και πρέπει να περάσουν από την εθνική κλίμακα στην ε, διεθνή. Πρέπει επίσης να δούμε ότι έχουν επίγνωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών τους ευθυνών οι νέοι αυτοί επιχειρηματίες. Η νέα αυτή γενιά χρειάζεται δημόσια στήριξη και με καινοτομία να δοθεί πρόσβαση σε πιστώσεις αυτές τις νεοσύστατες εταιρείε που είναι υπεύθυνε για τη δημιουργία περίπου 50% των θέσεων απασχόληση στην Ευρώπη. Οι εταιρείε που δημιουργήθηκαν μεταξύ 2008 και 2012 γνώρισαν ένα ποσοστό αποτυχία 40%. Οι δημόσιε πολιτικέ που στοχεύουν την οικονομική ανάπτυξη για τι επιχειρήσει και τον επιχειρηματικό κόσμο έχουν τώρα μια νέα πρόκληση μπροστά του. Την παρακολούθηση και την στήριξη τη επιβίωση αυτών των νέων εταιριών. Για να ολοκληρώσω, επιτρέψτε μου τον περασμένο μήνα μια από τις εταιρείες μας ε, κέρδισε σε ένα μεγαλύτερο διαγωνισμό νεοσύνθετων εταιρεών ε, ε, στην Ευρώπη. Μια εταιρεία της Startup Lisboa και επίσης το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, το LSE, έχει αναφερθεί πολλέ φορές θετικά για την startup Lisboa. Ε, δικός μας ρόλος και ο δικός μας καθημερινός αγώνας είναι να γίνει εφικτό ε, για μια εταιρεία του ψηφιακού κόσμου, να γίνει επιχείρηση και να πάρει ευρωπαϊκές διστάσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Βασκοσέλου Και τώρα ο λόγος στο δόκτορα Oliver Φρόμ του Unicastle Transfer. Απλώς να τονίσω και το εξής. Ε, θυμήσατε τον ρόλο των πανεπιστημίων. Μερικές φορές είναι, υπάρχουν και όρια στην ε, δυνατότητα δράσης των πανεπιστημίων και το πόσο μπορούν να συμβάλλουν στην δράση. Ίσως λοιπόν και ο κύριος Φρόμος ε, καθηγητής θα μπορούσε να μας ε, δώσει περισσότερα στοιχεία. Yeah, sehr Πρόεδρε, και αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω για το Πανεπιστήμιο του Κάσελ και τις δραστηριότητε του. Στο Πανεπιστήμιο του Κάσελ τα περασμένα χρόνια από την ε, κυβέρνηση της Γερμανίας ε, υπήρξε ένα βραβείο και είμαστε ηγετικοί στη Γερμανία. Να σας αναφέρω λοιπόν ποιες δομές και ποια μέτρα από πλευράς μας θεωρούμε ότι υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα από πλευράς των πανεπιστημίων και βοηθούν τα πανεπιστήμια. Αφενός θα ήθελα να σας παρουσιάσω πώς ε, μπορούμε να προωθήσουμε περισσότερο την ε, δημιουργία επιχειρήσεων από τα πανεπιστήμια και ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν κατά δεύτερον λόγο στην κοινωνία και την οικονομία που βασίζεται στη γνώση, ε, δημιουργούνται νέες επιχειρήσεις, είτε μέσω νέων επιχειρήσεων, με νέων προϊόντων, είτε μέσω νέων μοντέλων, εφίων μοντέλων επιχειρηματικότητας. Συχνά από τα πανεπιστήμια, γιατί είναι οι απόφοιτοι αυτοί που δημιουργούν ε, επιχειρήσεις και συχνά είναι αυτοί που φεύγουν από το σχολείται από τις σχολές αυτές που έχουν επιχειρηματικό πνεύμα. Είναι καθοριστικό λοιπόν τα πανεπιστήμια για τη δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ένα βασικό στοιχείο είναι το θέμα της επιχειρηματικότητας που αποτελεί τμήμα της στρατηγικής ανάπτυξης των πανεπιστημίων. Θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της ανάπτυξης των πανεπιστημίων. Πέρα από την ε, μεταφορά γνώσης, τη διδαχή, θα πρέπει και εδώ είναι σημαντικό ο τομέα τη μεταφορά γνώσεων, το τονίζω. Τα πανεπιστήμια το αναγνωρίζουν αυτό σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν έχει περάσει αυτό παντού. Ότι αυτή η πρόθεση τη ίδρυση επιχειρήσεων δεν είναι αντίθετη στην έρευνα και την ανάπτυξη. Αντιθέτω, γιατί υπάρχει στενή συνεργασία με τον επιστημονικό κλάδο. 98% στην ε, στο Κάσελ, 98% των επιχειρήσεων συνεργάζονται με τον μονοκατεμαϊκό κύκλο. Υπάρχει λοιπόν ένα βυσικό βιότοπο, όπου στηρίζει ο ένα τον άλλον. Θα πρέπει λοιπόν να πετύχουμε στην έρευνα συστηματικά να αναζητάτε και το δυναμικό εφαρμογής, να γίνει αυτό, αν θέλετε, το τμήμα τη νοοτροπία στα πανεπιστήμια. Είναι μια κουλτούρα λοιπόν ιδεών και επιχειρηματικότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει κάθε καθηγητής να ιδρύει μια εταιρεία. Όχι. Να μεταφέρει όμως την ιδέα αυτή. Η επιστήμη έχει και μία, ένα καθήκον τέτοιο, μία ευθύνη τέτοια. Γιατί στη τελική ανάλυση πολλά χρήματα δαπανώνται για τα πανεπιστήμια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σε ό,τι αφορά την έρευνα και κάθε ερευνητή θα πρέπει να αναζητά, να αναζητά πρακτικές εφαρμογές της έρευνάς του και μετά θα πρέπει να υπάρχουν και συστήματα υποστήριξης για την ε, εφαρμογή της ιδέας αυτής στη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο του Κάσελε σε όλες ε, τις κατευθύνσεις διδάσκουμε επιχειρηματικότητα όχι μόνο επιχειρηματικές γνώσεις, αλλά και η επιχειρηματικότητα, η νοοτροπία του επιχειρήν. Αυτό είναι πολύ πιο ευρύ πεδίο για να αναπτυχθούν ιδέες, έργα και να εφαρμοστούν στην πράξη. Αυτή η ικανότητα της επιχειρηματικής σκέψης δεν έχει εφαρμογή μόνο όταν ιδρύει κανείς μια επιχείρηση, αλλά και όταν εργάζεται σε μια επιχείρηση, σε μια οικονομία κοινωνική και οικονομική. Όλα αυτά λοιπόν μας επιτρέπουν να εκτιμούμε και τους κινδύνους. Σε αυτή την ε, ευρεία έννοια θεωρούμε ότι υπάρχει αποδοχή σε όλες τις σχολές και σε όλες τις κατευθύνσεις, γιατί είναι συχνά δύσκολο να βάλουμε ένα τέτοιο μάθημα σε καλλιτεχνικές σχολές. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό άρνησης, αλλά αν εξηγήσουμε ότι μετά το καλλιτέχνημα, το προϊόν θα πρέπει να διατεθεί στην αγορά, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αποδοχή. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε πάντα εξύπνα το πώς εντάσσονται οι η κλάδη αυτή στα πανεπιστήμια, γιατί θα πρέπει να συνάδει αυτό και να εναρμονίζεται με το βασικό ενδιαφέρον των επιστημόνων. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό αυτά τα θέματα να τα πραγματεύονται από μόνα τους στα πανεπιστήμια θεωρούμε ότι αυτά δεν θα πρέπει να τα επιβάλλουν τρίτοι, αλλά να τα αναπτύσσουν τα ίδια τα πανεπιστήμια. Αν υπάρχει ένα κέντρο του πανεπιστημίου, για παράδειγμα, στις πανεπιστημίου πόλης, αυτό αποτελεί ένα Αυτό σημαίνει ότι, αν παράδειγμα υπάρχει ένα κέντρο προώθησης επαγγελματικότητα, το οποίο φτιάχνει το ίδιο το πανεπιστήμιο, γίνεται πολύ πιο αποδεκτό ως συστατικό στοιχείο της ίδιας της σχολής. Και τώρα να περάσω στο δεύτερο τμήμα, στο ερώτημα του πώς το δυναμικό αυτό το οποίο έχουμε, αυτές οι ιδέες που έχουμε και προκύπτουν από την έρευνα και την ανάπτυξη, μπορούν να προωθηθούν πραγματικά. Υπάρχουν πανεπιστήμια, τα οποία, στα πανεπιστήμια μάλλον υπάρχουν δύο κίνδυνοι. Ο πρώτο κίνδυνο είναι να αναπτυχθεί κάτι το οποίο δεν χρειάζεται κανένας. Αυτός ε, ο κίνδυνος ε, υπάρχει για όλους, αλλά είναι πολύ έντονος στην επιστήμη. Ιδιαίτερω αν οι επιστήμονε κλείνονται στα δωματιάκια τους και δεν ε, ψάχνουν ποια είναι η σύνδεση με την πραγματική ζωή. Γι' αυτό λοιπόν είναι προτεραιότητα της προώθησης της επιχειρηματικότητας είναι προτεραιότητα να φροντίσουμε οι ιδέες ακόμα και όταν είναι πολύ ανώριμε σε πρώιμο στάδιο ακόμα, να έχουν επαφή με την πράξη, να υπάρχει ένα feedback από την πραγματική ζωή. Να μην ε, Χρειάζεται βέβαια να υπάρχει επιχειρηματικό σχέδιο. Να μπορεί κανείς, ε, αν έχει μία ιδέα, να ρωτήσει τον κόσμο αν του αρέσει. Πειραματικό λοιπόν έργο. Αυτό δούλεψε πολύ ε, καλά σε εμά. Όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο του Κάσελ, αυτή, η, αυτός ο ανταγωνισμός ε, ιδεών, αυτή η προώθηση ιδεών, όχι επιχειρηματικών σχεδίων, αλλά ιδεών. Όχι για να βρούμε ίσως την καλύτερη δυνατή ιδέα, δεν ξέρουμε ποια είναι η καλύτερη ιδέα, αλλά για να υπάρξει ε, δημοσιοποίηση, να γνωρίσει η κοινή γνώμη, οι επιχειρήσεις για παράδειγμα τις ιδέες αυτές. Το δεύτερο σημείο που είναι σημαντικό. Η επαφή των νέων με την ε, επιστήμη με τις ε, οικονομία, με τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, ε, η οικονομία βρίσκει ιδέες στο πανεπιστήμιο που την ενδιαφέρουν. Για τους ε, νέους φοιτητές και επιστήμονες πρόκειται για τους πρώτους χρηματοδότες και έτσι λοιπόν μπορεί να δημιουργηθεί ένα δίκτυο αμοιβαίας υποστήριξης. Έχουμε λοιπόν στο Κάσελε ένα συμβούλιο επιχειρηματιών και εδώ οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, να οικοδομήσουν δίκτυα και να ακούσουν κάποιες πρώτες εντυπώσεις. Πέρα από τον κίνδυνο της αγοράς υπάρχει και ο κίνδυνος της χρηματοδότησης ασφαλώς. Πολλά ακούσαμε για αυτό το θέμα σήμερα. Γι' αυτό δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να τα επαναλάβω, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ένα σημείο το οποίο και αναφέρθηκε στο προηγούμενο πάνελ, το crowdfunding πρόκειται για ένα εξαιρετικό εργαλείο για ομάδες σε πολύ πρώιμη φάση. Σήμερα θεωρώ ότι η χρηματοδότηση ε, έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση έργων, όχι με επενδύσεις, που και αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο. Γιατί έτσι δεν δημιουργούνται μόνο χρήματα, αλλά υπάρχει και επαφή με την αγορά. Πολύ χρήσιμη λοιπόν ιδέα. Τα έργα μας λοιπόν έχουν να κάνουν με την προχρηματοδότηση των προϊόντων, δηλαδή ε, πολλούνται προϊόντα προτού παραχθούν μεταξύ 50 και 100.000 ε, ευρώ. Είμαστε λοιπόν το πρώτο πανεπιστήμιο που έχει δημιουργήσει μια τέτοια πλατφόρμα. Αυτό λοιπόν καλύπτει ένα κενό και επιτρέπει και τη μετέπειτα χρηματοδότηση. εφόσον ο κόσμος δηλαδή ε, ήταν σε θέση και ήταν τεθειμένος να πληρώσει για προϊόντα που δεν υπήρχαν ακόμα. Είναι λοιπόν εξαιρετικό το εργαλείο αυτό και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε από την πολιτική να μην το περικόψει. Και θα ήθελα να κλείσω λοιπόν με αυτά και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε για αυτήν την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Η τελευταία παρέμβαση κυρία Κάρλα Φανστίνμπεργεν, υπεύθυνη νομικών θεμάτων του Materialize. Um, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Φιλίπ Ντεμπάκερ για να... γιατί με κάλεσε να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία που είχαμε με μια βελγική καινοτόμος εταιρεία, η οποία ε, η Materialize λοιπόν είναι μια βελγική εταιρεία αρχικά, ιδρύθηκε το 1990. Αυτή είναι η φωτογραφία του ιδιοκτήτη. Ξεκίνησε την εταιρεία με φίλους του από το Πανεπιστήμιο. Έχει μεγαλώσει αρκετά η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο βάσει του δίκτυ Nasdaq ε, φέτος. Έχουμε ξεπεράσει πλέον τα μεγέθη της μικρομεσαίας επιχείρησης. Αυτό όμως δεν αλλάζει και τίποτα σημαντικό. Είμαστε επιχειρηματική εταιρεία. Μας αρέσει να καταπιανόμαστε δηλαδή με πράγματα. Θέλουμε να ε, ε, επινοούμε νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα, να διερευνούμε, να φτάνουμε την τεχνολογία στα άκρα της, να την ε, διερευνούμε μέχρι τέλους και θέλουμε να έχουμε ε, τεχνολογική καινοτομία. Η Materialize είναι δραστήρια στην τρισδιάστατη εκτύπωση. Βλέπετε εδώ ένα δείγμα εκτύπωση σε τρεις διαστάσεις ενός ιατρικού μοντέλου ε, στη δεκαετία του 1990. Βλέπετε αυτή την πολύ αδρή επιφάνεια η οποία τότε χρησιμεύε ιδιαίτερο στους χειρουργούς και στους κλινικούς ερευνητές για να βελτιώνουν τη θεραπεία που προσέφεραν στους ασθενείς τους χάρη στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίσαμε να βελτιώνουμε την τεχνολογία μας και μπορούμε να εκτυπώσουμε αντικείμενα όπως αυτό που βλέπετε εδώ, ε, βάσει των δεδομένων ιατρικής απεικόνησης. Και αυτό είναι ε, δοκιμαστικό για τους ε, ε, χειρουργούς αλλά και για το σχεδιασμό του εμφυτεύματος το οποίο θα υλοποιηθεί τελικά για να ε, καλύψει ελλείμματα των ασθενών τα οποία έχουν προκληθεί από μια πλειάδα παθήσεων. Πριν μπω στα θέματα έρευνας και ανάπτυξης, θα ήθελα να σας δείξω αυτό εδώ το παράδειγμα. Ακουστικά βοηθήματα, διάφορα ακουστικά βοηθήματα βλέπετε στην εικόνα, την περασμένη ε, δεκαετία Πρέπει να ξέρετε ότι τα ακουστικά βοηθήματα σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον δεν παράγονται κλασικά, αλλά εκτυπώνονται με την τρισδιάστατη εκτύπωση. Η έρευνα λοιπόν και η ανάπτυξη είναι καθοριστική για την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Μέρος του κύκλου εργασιών μας τον επενδύουμε συνεχώς. Δεν το χρηματοδοτούμε εμείς μόνο αποκλειστικά. Πάρα πολλά κονδύλια έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχουμε σε διάφορα ερευνητικά έργα. Και αυτό μας έχει βοηθήσει να καταλήξουμε σε πολύ σημαντικές τεχνολογικές ε, εφαρμογές. Βλέπετε λοιπόν την τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ένας τρόπος κατασκευής ε, προϊόντων ο οποίος λειτουργεί αντίθετα από ότι ο κλασικός. Χτίζουμε ένα προϊόν στη βάδα αναστιβάδα, προσθέτουμε υλικό παραγωγή στο προϊόν και σιγά σιγά αυτό αναδύεται από τον εκτυπωτή. ενώ στην παραδοσιακή κατασκευή αφαιρούνται υλικά έτσι ώστε να σμιλευτεί το προϊόν στο σχήμα ε, που, θέλει κανείς. Πολλοί κόσμος πιστεύει ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση σημαίνει ότι θα αγοράσω ένα μηχάνημα, θα πατήσω ένα κουμπί και θα βγει ένα προϊόν. Ε, σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό. το μηχάνημα θα τυπώσει αυτό που ε, το τροφοδοτήσετε. Αν το τροφοδοτήσετε με ε, σκουπίδια, σκουπίδια θα, βγουν από το μηχάνημα. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό να επενδύει κανείς στην αγορά μηχανομάτων, αυτό μας λέει ο διοκτήτης, τα εγκατέστησα, προσέλαβα τους ανθρώπους και άρχισα να παράγω. Είναι ένας από τους τρόπους αυτός. Να ξεκινήσει κανείς να είναι δραστήριος στον κλάδο της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Δεν είναι όμως ο μόνος. Με την ψηφιοποίηση της οικονομίας Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες. Μπορεί κανείς να χτίσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα και εκεί να ανοίξει το δρόμο στους σχεδιαστές, να ε, φορτώσουν αυτή τα σχέδιά τους, να τα εκτυπώσει κανείς και να τους τα παραδώσει και έτσι αρχίζουν και δημιουργούνται νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και δημιουργούνται νέες επιχειρήσεις. Πελάτες της δικής μας διαδικτυακής πλατφόρμας που μας είχαν αναθέσει να εκτυπώσουμε τα προϊόντα τους, ε, ξανάρχονται και δεν θέλουν πια να τα εκτυπώσουμε ε, για τον εαυτό τους, για τους φίλους τους, για τις οικογένειές τους, αλλά μας ε, δίνουν παραγγελία για βιομηχανική εκτύπωση γιατί έχουν να τα πουλήσουν σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Βλέπετε λοιπόν ότι τι μπορώ να κάνω με αυτή τη διαδικτυακή πλατφόρμα την οποία ε, έχω στη διάθεσή μου. Είτε ασχολούμαστε με τις ιατρικές εφαρμογές, είτε με τις ε, τεχνολογικές εφαρμογές, είτε με σχέσεις επιχειρήσεων προς ε, καταναλωτές, η ποιότητα βρίσκεται στο κέντρο. Στο επίκεντρο όλων αυτών που κάνουμε, όπως βλέπετε, είναι μια σχετικά νέα τεχνολογία, υπάρχουν κάποιες ε, αστοχίες αν θέλετε, υπάρχουν κάποιες παγίδες να το πω έτσι, δεν τις έχουμε ξεπεράσει όλες, όμως ανεξαρτήτως όλων αυτών και των προκλήσεων που υψώνονται μπροστά μας, το βασικό μέλημα για μας είναι η υψηλή ποιότητα των προϊόντων. Να παραδίδουμε στους πελάτες μας ε, προϊόντα πραγματικά υψηλής ποιότητας. Θα ήθελα κάποια στιγμή, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας μιλήσω για τις προκλήσεις. Η Materialize, η εταιρεία μας, δεν θέλει μόνο να έχει επιτυχία, αλλά θέλει να είναι και το λίκνο των νέων ιδεών. Σε εμάς θέλουμε να ε, δημιουργείται οτιδήποτε νέο. Δεν μιλώ και βέβαια σε αυτό υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι οι νομοθετικές αλλαγές. Με την τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί κανείς να εκτυπώσει οποιοδήποτε σχέδιο, να κάνει σάρωση ενός προϊόντος, να κάνει αντίστροφη μηχανική αυτού του προϊόντος, να φτιάξει φάκελο και να εκτυπώσει αυτό το φάκελο. Βλέπετε αυτό το κύβο, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί μάλιστα και σε ταινίες και είχαμε είχαμε ε, την πρώτη νομική διαμάχη με τον σχεδιαστή, ε, με έναν σχεδιαστή που διεκδικούσε ότι είχε φτιάξει εκείνο αυτό, το τον κύβο, τον Super 8. Σε κάθε περίπτωση Υπάρχουν θέματα ε, παραβάσεων του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, ε, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ούτω καθεξής. Ε, αυτά πρέπει να τα δούμε. Εδώ βλέπετε χειρουργικούς οδηγούς. Είναι ένα προϊόν που εκτυπώνεται σε τρεις διαστάσεις με βάση την απεικόνιση την ιατρική των δεδομένων των ασθενών είναι ένα τεράστιο βοήθημα για το χειρουργό που ε, κάνει ορθοπαιδική χειρουργική χειρουργεί ένα ε, οστούν που έχει κάταγμα και μπορεί έτσι να διασφαλίσει ότι το μέγεθος του εμφυτεύματος που θα χρησιμοποιήσει είναι το σωστό. και έτσι περιορίζεται ο χρόνος στο χειρουργικό τραπέζι είναι ε, μικρότερος ο χρόνος ανάρρωσης και χαμηλότερος ο κίνδυνος φλεγμονής. Σε κάθε περίπτωση έχουμε το νέο σχέδιο κανονισμού για τις ιατρικές συσκευές και εξαρτήματα Υπάρχουν διάφορες διατάξεις για τις ιατρικές συσκευές που κατασκευάζονται ή το χύψη ιατρικό εξάρτημα που κατασκευάζεται για τις ανάγκες συγκεκριμένου ασθενούς και θεωρούμε ότι θα υπάρξει πρόβλημα, έχουμε καθυστέρηση, ε, ενώ μία άλλη πρόκληση είναι η εξής. Για την τρισδιάστατη εκτύπωση πρέπει να αναθεωρήσουμε εκ βάθρων την έννοια του customization, του, προσαρμόζω κάτι στις ανάγκες της συγκεκριμένης του εκάστοτε πελάτη. Ε, υπάρχει τεράστια προστιθέμενη αξία σε ασθενείς με ε, πολύ σπάνιες νόσους και... Πρέπει να πούμε ότι για ότι είναι πολύ δύσκολο να έχουν πρόσβαση στην αγορά πάρα πολλά ιατρικά εξαρτήματα ή συσκευές τα οποία είναι σπάνια ή χρησιμοποιούνται για σπάνιες περιπτώσεις. Ε, με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις. Αν κανείς συγχρηματοδοτήσει την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας χωρίς τη συνέχεια να παρέχει το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να τεθούν σε εμπορία αυτά τα νέα προϊόντα που έχουν επινοήσει οι εταιρείε, ε, τότε είναι κρίμα ο κόπος του και τα λεφτά που έδωσε εξ αρχής. Νομίζουμε ότι μπορεί να υπάρχει πραγματικά ε, σημαντική προστιθέμενη αξία. Το εμφύτευμα που σας δείχνω εδώ εκτυπώθηκε μέσα σε 5 ώρες. Σχεδιάστηκε όμως μέσα σε 95 ώρες. Είναι μια τεχνολογία η οποία χρηματοδοτήθηκε για έξι ολόκληρα χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Λουβέν ε, σε συνεργασία με τη δική μας εταιρεία την Materialize. Έχουμε βοηθήσει 100 ασθενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το ε, προϊόν, με αυτό το εμφύτευμα και τώρα ο νόμος αλλά και η κοινωνική ασφάλιση απαγορεύει τη θέση σε εμπορία γιατί υπάρχει ένας περιορισμός της τιμής ο οποίος ε, είναι τελείως ασύμφορος για μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το παράγουμε. Και ακόμα και αν ξεπεράσουμε τους περιορισμούς της βελγικής νομοθεσίας, τότε θα πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία σε κάθε χώρα μέλος και δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Είναι κρίμα. Θα πρέπει να υπάρχει τρόπος να λυθεί αυτό το ζήτημα νομικά. Από εκεί και πέρα. Έχουμε και βιομηχανικές εφαρμογές Το είπα και πριν. Ευθύνη του κατασκευαστή, εάν συνεχίσουμε να τα πουλάμε. Αυτά λοιπόν με τις βασικές προκλήσεις, νομίζω τέσσερις ανέφερα τελικά, ε, αυτά είχα να πω προς το παρόν στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Καταγράφουμε το σχολείό σας για τη νομοθεσία για τα, για τα ιατροτεχνολογικά, αλλά το σημειώνουμε. Δεν είναι αυτό βέβαια το θέμα μας, αλλά ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και η ενεξελίξη αναθεώρηση. Και τώρα ο λόγος στον συνάδελφο Ντεμπάκερ για την πρώτη παρέμβαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους τρεις ομιλητές για τις μαρτυρίες τους. Νομίζω ότι αυτό που γίνεται σαφές από τις ε, παρουσιάσεις σας και ο λόγος που είχαμε και την ακρόαση σήμερα το πρωί είναι ότι θέλαμε να μάθουμε τις απόψεις όσων καθημερινά ασχολούνται με τα θέματα αυτά και να δούμε πώς χειρίζεσαι την νομοθεσία από την αντίθετη προοπτική από τη δική μας, από τις μαρτυρίες σα, νομίζω έγινε σαφέ ότι ενώ μπορούμε να καλύψουμε όσο περισσότερα στοιχεία μπορούμε και ενώ προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη το ρόλο των νεοσύστατων επιχειρήσεων, τελικά δεν είμαστε πάντοτε τόσο επιτυχείς. Γι' αυτό έχω μια σειρά από ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα, για τα νομοθετικά κείμενα βλέπουμε ότι η Ευρώπη δεν καταφέρνει να μετατρέψει τα διπλώματα βρεσιτεχνία σε προϊόντα, όπως επιτυχημένα κάνουν άλλες ε, περιοχές. Ε, πρωτοβουλίες υπάρχουν από κέντρα, πανεπιστήμια, με ολόκληρες, ε, ολόκληρα τμήματα και μια σειρά από ανθρώπους για να βοηθήσουν εδώ, αλλά δεν τα καταφέρνουν πάντοτε. Και σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο η δράση δεν είναι ακόμα αρκετή. Πιστεύετε εσείς ότι θα πρέπει τα πράγματα να παραμένουν όσο έχουν κοντά στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ε, ιδρύματα ή ότι θα πρέπει να φτιάξουμε δίκτυα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερη ερώτηση. Κάτι που και εσείς το υπενηθήκατε, ότι όταν θέλει κανείς να εμπορευτεί ένα προϊόν, στην εσωτερική αγορά της Ευρώπης δεν υπάρχει πλήρης ολοκληρωσία. Αυτό μας απασχολεί και εμάς πολύ. Και σήμερα με την κρίση βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν τάσεις προστατευτισμού αντί να απελευθερώνουν την αγορά τους. Αυτό ως Επιτροπή Τρέ θα πρέπει να το έχουμε κι εμείς υπόψη. Και μια τελευταία παρατήρηση, γιατί θα ήθελα μετά να ε, προλάβω να ακούσω και απαντήσεις. Ε, έχετε ασχοληθεί με τα προγράμματα που αφορούν, έχετε δει όλη την διαδικασία μάλλον από τη φάση ίδρυσης μιας μικρομεσαίας μέχρι τη φάση που εισάγεται στο χρηματιστήριο. Ε, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόσβαση στις πιστώσεις, ε, στην λειτουργία σας στην αγορά, ήταν στην αρχή ή όταν η εταιρεία ορίμασε. Ε, τις δυσκολίες πώς θα τις περιγράφατε μέσα από τις φάσεις της ορίμανσης. Πού ήταν τα πιο δύσκολα, στην ε, αρχή, στη μέση, στην ορίμανση. Ευχαριστούμε η κυρία Κάλλας. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Μία ερώτηση έχω να κάνω σε ό,τι αφορά μια νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συζητιέται εδώ. Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά απόρριτα και την προστασία τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει στην μελέτη Τύπου ότι είναι υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ε, νεοσύστατων εταιριών, καθώς δεν έχουν αρκετά χρήματα να καλύψουν τα απορριτά τους με ε, διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Συμφωνείτε με τις απόψεις αυτές. Ή πιστεύετε ότι τέτοιου είδους προστασία εμπορικών απορρίτων μπορεί να δημιουργήσει φράγματα, προσκόμματα στην αγορά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Ο κ. Γκρομπατσίτς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, στον κύριο Βασκόνσης. Στα πλαίσια της πρόθεσης της επιχειρηματικότητας που ζητάτε και με το οποίο ασχολείστε στη Λισαβόνα. Πείτε μας. Είπατε ότι οι νέοι δεν θέλουν να ιδρύσουν δικές τους εταιρείε για μια σειρά διαφορετικών λόγων, τους οποίους και αναφέρατε. Ένας εξ αυτούς είναι οι χαμηλές αποδοχές. Φυσικά οι αποδοχές δεν είναι θέμα γιατί δεν είναι το θέμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι ερμήνευσα τα λόγια σας. Πείτε μας, ίσως, τι πιστεύετε. Ποιοι είναι οι λόγοι για την έλλειψη ανάπτυξης, την έλλειψη ευκαιριών για τις ε, νεοσύστατες εταιρείες. Και μία ερώτηση έχω να κάνω στον Dr. Φρόμ. Ε, είπατε ότι ολοκληρώνεται μία περίοδος όπου οι ερευνητές θα πρέπει να καταρτήσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο και να αποφασίσουν πώς θα αναπτύξουν οι ίδιοι τις επιχειρήσεις τους. Πείτε μας λοιπόν, πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να δημορφωθεί σήμερα ο ρόλος των επιστημόνων στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και τελευταία ερώτηση προς την κυρία Στάνμπεργκ. Όταν αναπτύσσει κανείς την επιχείρησή του, πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει πιο πολύ ή πιο λίγη νομοθεσία από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. για να αποφύγουμε τους περιορισμούς που επιβάλλει η ρύθμιση και η νομοθεσία. Πείτε μας λοιπόν την απόψή σας ως επιχειρηματίας από αυτόν. Ευχαριστούμε. Τελευταία παρέμβαση ο συνάδελφος Ζωρίνιου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα μιλήσω τη μετρική μου γλώσσα. Να ευχαριστήσω τους ε, παρεμβαίνοντες. Όλες οι ομιλίες μας έδωσαν ελπίδες για το μέλλον και φαίνεται να ανοίγουν το δρόμο ε, για να μπορέσει να αναλάβει ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση στο νέο κύκλο ψηφιοποίηση σε παγκόσμια κλίμακα, παρόλο που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Startup Lisboa έχει μια διπλή ιδιότητα. Ε, στηρίζει επιχειρηματίες αλλά ταυτόχρονα και η ίδια είναι ε, επιχειρηματική, έχει επιχειρηματική διάτρωση δηλαδή έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο, ένα franchise αυτής της φιλοσοφίας της σε άλλες πόλεις, σε άλλες πόλεις της Πορτογαλίας. Νομίζω ότι σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς τέτοια δίκτυα θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ συχνά λέω ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να δώσει τέρμα στους φορολογικούς παραδείσους και για κάθε φορολογικό παράδεισο που θα πάψει να υπάρξει θα έπρεπε να υπάρχουν 100 επενδυτικοί παράδεισοι ε, αντιστοίχως. Τι περιμένουμε ε, λοιπόν, ε, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι περιμένετε από την πλευρά των πολιτικών ηθινόντων, τι νομοθετικές πρωτοβουλίες, τι κίνητρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξει αυτά τα δίκτυα, διότι τα δίκτυα αυτά είναι ε, ουσιαστικής σημασίας. Τι στήριξη θέλετε, τι λείπει για σας, κατά την άποψή σας. Αυτό πρέπει να ξέρουμε από αυτήν την ακρόαση, πιστεύω. Ε, και πάλι μπράβο σε όλου. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Δεν υπάρχουν άλλε παρεμβάσει. Να έχουμε ένα τελικό γύρο απαντήσεων. Να, να παρακαλέσω να παραμένετε στα τρία λεπτά ο καθένα από του παρεμβαίνοντε. Και προσπαθήστε να απαντήσετε όσο δυνατόν ακριβέστερα. Πρώτο ο κ. Βασκονσέλου. να απαντήσω στην ερώτησή σας για τα φράγματα, τους φραγμούς στην επιχειρηματικότητα. Από την δική μου την πείρα και επειδή τον κόσμο των επιχειρήσεων τον παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια, Έχω, υπάρχουν χιλιάδες λόγοι. Αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε και εκεί πρέπει να παρέμβουμε και να αλλάξουμε τα πράγματα Προφανώ δεν θα είναι το επίπεδο τη νοοτροπία, ούτε των κοινωνικών επιστημών, ούτε τη αντίληψη του κινδύνου των αποτυχιών. Αυτό που εμεί μπορούμε να κάνουμε και εσεί ω νομοθέτε και ω πολιτικοί θύνοντε είναι να κάνουμε κάτι στη νομοθεσία για την πρόσβαση στις πιστώσεις, για την φάση ίδρυσης μιας επιχειρήσης. Και ακόμη πιο σημαντικό, στην Πορτογαλία ή κι αλλού, ε, στο, στη φάση κλεισίματος μιας επιχείρησης που και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην Ευρώπη. Ο τρόπος που κανείς αναγκάζεται να σταματήσει την εμπορική του δραστηριότητα τον εμποδίζει να συνεχίσει με κάτι διαφορετικό. Είμαστε λοιπόν εδώ γρήγορα αποτελέσματα. Και ε, ίσως κάτι που δεν ξέρετε είναι ότι στη Λισαβόνα, στην Πορτογαλία τα αποτελέσματά μας μπορεί να λειτουργούν ε, να έχουν επιτευχθεί πάρα πολύ γρήγορα, αλλά έχουμε διάρκεια, ε, έχουμε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Συνεργαζόμαστε με πανεπιστημιακά κέντρα και για πρώτη φορά έρχονται πιο κοντά στον επιχειρηματικό κόσμο. Για πρώτη φορά λένε στους νέους που φιλοδοξούν να δουλέψουν σε μεγάλες επιχειρήσεις ότι υπάρχει λύση να φτιάξουν τη δική τους εταιρεία. Να δώσουν σάρκα και οστά στα όνειρά τους χωρίς να κάθονται μια ζωή να υλοποιούν όνειρα άλλων. Τρία χρόνια πριν Εάν ήμουν σε μια τάξη πανεπιστημίου στη Λισαβόνα, σε ένα αμφιθέατρο και ρώταγα τους νέους πόσοι θα ήθελαν να γίνουν επιχειρηματίε, 4-5 θα σήκωναν το χέρι. Τώρα είναι πολύ περισσότεροι. Στη δική μου τη γενιά, στη Λισαβόνα, η φιλοδοξία όλων ήταν να δουλέψουν για τι χρηματοπιστωτικέ αγορέ, για την Goldman Sachs, για το City στο Λονδίνο ή τη Wall Street στη Νέα Υόρκη. Τα πράγματα έχουν ανάξει. Ε, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ε, τώρα είναι η στιγμή να έχουμε νέους επιχειρήσεις. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ζωρίνιου όλες για την ερώτησή του. Όντα, όντως, σε συνεργασία με το Δήμο της Λισαβόνας ε, ιδρυθήκαμε και ε, με άλλες επιχειρήσεις που μας στήριξαν έχουμε περάσει ήδη στο Πόρτο και σε άλλες μεγάλες πορτογαλικές πόλεις. Πάντω να πω ότι η Startup Lisboa για την ώρα δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από κοινοτικά κονδύλια, ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από κανένα δημόσιο ταμείο. Για πολλούς λόγους, αλλά γιατί ήδη η Λισαβόνα δεν βρίσκεται στις περιοχέ σύγκληση και δεν έχει δικαίωμα στήριξη. Λισαβόνα, να το πω για όσους δεν το ξέρουν, είναι το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό κέντρο της Πορτογαλίας. Είναι το μέρος όπου υπάρχουν περισσότεροι ερευνητές, όπου υπάρχουν, ε, υπάρχει επιστημονική γνώση, περισσότερο δυναμικό για τεχνολογικούς, για επιχειρηματίες στον χώρο της τεχνολογίας. Υπάρχουν περισσότεροι ερευνητέ και δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ για να στηριχθούν οι νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται εκεί. Εάν εδώ μπορούσατε κάτι να κάνετε, αυτή θα ήταν η τεράστια συμβολή για την δημιουργία θέσεων εργασίας και για να, παραμείνει, ε, στην, να παραμείνουν στην Πορτογαλία και στην Ευρώπη τόσες ε, επιχειρηματικές διάνοιες που αλλιώς θα διαφύγουν. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και τώρα κύριος Φρόμ. Δόκτορα Φρόμ. Ρωτήσατε Ποιε είναι οι δυσκολίε στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνία και την προστασία προϊόντων και διαδικασιών. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνία των πανεπιστημίων κατά κανόνα απέχουν πολύ από την αγορά και υπάρχει μεγάλη ανάγκη επαληθευσή τους για να καταδείξουμε ότι όντω λειτουργεί μια εφεύρεση σε ό,τι αφορά τα πρωτότυπα, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία προϊόντων και την διάθεση ενός προϊόντος το οποίο πραγματικά μπορεί να ε, εμπορευθεί. Βλέπουμε στα γερμανικά πανεπιστήμια τουλάχιστον ότι δεν υπάρχει τέτοια χρηματοδότηση. Δεν λαμβάνουμε χρήματα από το κράτο για τα θέματα αυτά. Και κατά δεύτερον, οι επιστήμονε δεν έχουν τι ικανότητε για να αναπτύσσουν τέτοια έργα. Μεταξύ ενός ε, έργου έρευνα το οποίο έχει ανοιχτό αποτέλεσμα και ενός έργου επαλήθευση στην αγορά που ορίζεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο με το οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε προκειμένου να αναπτυχθεί ένα προϊόν για την αγορά υπάρχει μεγάλη απόσταση. Πρόκειται για δύο διαφορετικά τελείως πεδία και δεν έχει να κάνει αυτό τίποτα με την δραστηριότητα των επιστήμονων. Χρειαζόμαστε δηλαδή και χρηματοδότηση, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά μεθοδολογία για τους, επι... για τους επιστήμονες. Δεν μπορούν να υποστηρίξουν τα θέματα αυτά, δεν είναι το τομέα τους. Υποστήριξη λοιπόν μεθοδολογική. Και αυτό ε, φέρνει μεγάλο βάρος στα πανεπιστήμια γιατί είναι μεγάλη ανάληψη κινδύνου. Στην Γερμανία λοιπόν υπάρχει πρόσφατα προβλέφθηκαν κορβανάδας για το θέμα αυτό, αλλά αυτό αποτελεί και ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ξεχωριστή λοιπόν προώθηση της επαλήθευση, εξακρίβωσης των προϊόντων. Αυτό εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχει. Τώρα, για το θέμα των προσκομμάτων, των εμποδίων από πλευρά των πανεπιστημίων, μία βασική αρχή είναι ότι πρόκειται για θέμα προσωπικότητας, το θέμα του κατά πόσον οι επιστήμονε ε, φοιτητέ, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα μπορούν να εκπληρώσουν το ρόλο του επιχειρηματία. Αυτό το παρακολουθούμε πάντα με ενδιαφέρον. Μετά από έξι μήνες έρχεται ένας επιστήμονας, ένας φοιτητής και βλέπουμε ότι ενδεχομένως δεν είναι ένας καινούριος άνθρωπος. Αν υπάρχει λοιπόν αυτή η στάση, αυτή η προθυμία, αυτή η πίστη στο έργο, πολλά από τα προσκόμματα, πολλά από τα εμπόδια τα οποία πάντα ανακύπτουν, μπορούν να ξεπεριαστούν και είναι διαφορετικό αυτό ένα έργο. Δεν μπορώ να δώσω μία απάντηση που να ισχύει για όλα. Και εδώ λοιπόν είναι σημαντική η καθοδήγηση των έργων για τον ρόλο των επιστήμονων τώρα. Νομίζω ότι υπήρξε μία παρανόηση. Οι επιστήμονες θα πρέπει τουλάχιστον να είναι μέντορες των έργων αυτών, θα πρέπει να τα συνοδεύουν θετικά, αλλά φυσικά και μπορούν να συμμετέχουν ως μέτοχοι σε τέτοια έργα. Τέλος, πιστεύω ότι η μεταρρύθμιση δημιουργεί ένα πάρα πολύ σωστό πλαίσιο για τα πανεπιστήμια της Γερμανίας και στο Κάσελ συμμετείχαμε. Αυτό προϋποθέτει φυσικά ότι το Πανεπιστήμιο είναι προτίθεται να κινητοποιήσει τα μέσα συγχρηματοδότησης. Ε, Ευχαριστούμε. Τελευταία παρέμβαση. Η κυρία Κάρλα Φαν Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ως προς την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και για το κατά πόσο είναι πιο εύκολο για μια μικρή ή για μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Μπορώ να σας πω ότι είναι δύσκολο να πει κανείς ότι το ένα είναι πιο δύσκολο απ' τα άλλο. Οι διαφορετικές εμπειρίες είναι αυτό που ακριβώς που εννοώ, διαφορετικές. Δεν έχουμε αρχείο επιδόσεων για να αποδείξουμε αυτό που χρειάζεται και για να έχουμε δείξει στους επενδυτές ότι θα έχουν απόδοση στην επένδυση που θα κάνουν και αυτό είναι πρόβλημα. Τώρα, Δεν πρέπει τόσο να ασχολούμαστε με τα άλλα, όσο το να δείξουμε ότι δεν είναι σημαντικό ο επενδυτής μόνο να σκέφτεται την απόδοσή του σε βραχυπρόθεσμο ε, διάστημα. Όταν κάποιος, μια επιχείρηση κάνει τεχνολογία, φτιάχνει τεχνολογία, χρειάζεται επένδυση σε βάθος χρόνου, χρειάζεται επιμέλεια για να έχει πραγματικά την προστιθέμενη αξία. Δεν γίνονται όλα αυτά σε μία νύχτα. Από την άλλη το χρήμα δεν είναι τζάμπα. Αυτό είναι σαφέστατο. Και οι επενδυτές έρχονται να επιδίσουν με βάση το αρχείο επιδόσεων της εταιρείας τα τελευταία 20 χρόνια. Θα αρχίσουν να πιέζουν και θέλουν γρήγορα να δουν αποτελέσματα. Και θα πρέπει η επιχείρηση να ανταπεξέλθει και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει. Δεν λέω λοιπόν ότι το, η μία επιχείρηση έχει πιο εύκολο δρόμο στη χρηματοδότηση από ότι μια άλλη. Είναι απλά διαφορετικά. Κάθε φορά. Κατά τη γνώμη μας η ταυτότητα της επιχείρησης είναι εξαιρετικά σημαντική. Υπάρχει το μεγάλο εμπόδιο του να φτιάξει κανείς το χαρτοφυλάκιό του με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις πατέντα, πατέντες του. Ωστόσο, αν διαλέξει να πατεντάρει ορισμένα είδη τεχνολογίας, σίγουρα ε, θα πρέπει να δεχθεί ότι κάποια στιγμή η τεχνολογία αυτή θα μαθευτεί και θα είναι ανοιχτή, θα υπάρχει. Είναι όλο και πιο δύσκολο να έχει κανείς δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Φαινόμενα τύπου big data ε, θα οξύνουν αυτή τη δυσκολία και αυτό θα επηρεάσει τις μικρές επιχειρήσεις και τις μεγάλες. Θα πρέπει να αναθεωρήσουν ε, τη στρατηγική τους για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Θέλουμε δηλαδή να επενδύουμε συνεχώς σε εταιρείε που να πατεντάρουν τα πάντα και τελικά να επενδύουμε για τη δημιουργία μονοπωλίων. Από την άλλη, τα προβλήματα του να τα ανοίγουμε όλα και να τα έχουμε όλα διαθέσιμα είναι γνωστά. Χρειάζεται τώρα περισσότερη νομοθεσία ή αφαίρεση ε, κουραστικών και περιττών νομοθετικών διατάξεων. Δεν μπορώ να σας απαντήσω με σαφήνεια. Όταν έχουμε να κάνουμε με θέματα ένομης τάξης, π.χ. την ασφάλεια του ασθενούς, κανείς δεν αφισβητεί το ότι είναι ανάγκη ε, ο νόμος να είναι σαφής, αυστηρός και να ισχύει για όλους. Από την άλλη, δεν είναι δίκαιο ένας εργοδότης δύο υπαλλήλων να πρέπει να συμπληρώσει 40 έντυπα για να προσλάβει ένα τρίτο υπάλληλο. Και αυτό αλήθεια είναι. Πρέπει λοιπόν οι νομοθέτες να υιοθετούν νομοθεσία όπου θα προστατεύουν την ένωμη τάξη αλλά να μην υπερρυθμίζουν και νομοθετικά να προβλέπουν τα πάντα τα πάντα, γιατί ιδαλλιώς ουσιαστικά ποδοπατούν τις φιλοδοξίες του επιχειρηματία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ ε, και ευχαριστώ που σεβαστήκατε κατά χρονικά όρια. Στο κλείσιμο αυτής της πρωινής ακρόασης να ρωτήσω τον κύριο Ντεμπάκερ αν θέλει να κάνει κάποιες καταληκτήριες παρατηρήσεις. Έχετε ένα λεπτό για τα συμπεράσματα, εφόσον θέλετε. Παρακαλώ. Θα είμαι πολύ σύντομος, διότι πιστεύω ότι οι συμμετέχοντες των τριών διαφορετικών πάνελ μύρισαν τόσο καλά επικοδομητικά και με τόσο σαφή μηνύματα Ακούσαμε ποιο είναι ο ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την οικονομία, ακούσαμε πώ τι ε, εμποδίζουν στη λειτουργία του περίπλοκε νομοθεσίε και ευρωπαϊκέ αλλά και κατακαιρματισμό σε εθνικό επίπεδο τη νομοθεσία και είδαμε και τι σημαντικό ρόλο οι ιδιωτικοί επενδυτέ μπορούν να διδαματίσουν στην κινητοποίηση της οικονομίας, με τα κεφάλαια κινδύνου προς τις ε, καινοτόμες επιχειρήσεις και μάλιστα με γρήγορες ταχύτητες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις διαρκείας, όχι απλώς βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα για να χτίσουμε τις αυριανές μεγάλες επιχειρήσεις της Ευρώπης. Το τελευταίο πάνελ νομίζω ότι ήταν σαφές ότι η μεταφορά τεχνολογίας είναι ζωτική σημασία και επιτρέπει στις εταιρείε να χρησιμοποιήσουν την πιο πρόσφατη τεχνολογία εκνής στην έρευνά τους και να φέρουν αποτελέσματα χωρίς να εμποδίζονται πρέον από την ε, νομοθεσία συμβάλλοντα την αύξηση της αγοράς. Αυτά ήταν τα γρήγορα συμπεράσματα μου από τη σημερινή ακρόαση. Φυσικά στην έκθεση για την πράσινη οικονομία και την οικονομία των μικρομεσαίων θα ε, καταγράψουμε όλες αυτές τις παρατηρήσεις και θα φροντίσουμε να έχουμε γρήγορα μια έκθεση ώστε να ε, συμβάλλουμε και εμεί στην οικοδόμηση μιας ε, καλή αγορά για τις μικρομεσαίες σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονε και θα συναντηθούμε και πάλι στις 3.